Uh, ladies and gentlemen, uh, first of all, my apologies for being. Uh, Συγγνώμη που καθυστέρησα λιγάκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, στις 15 Φεβρουαρίου την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε χώρα ένα πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στο Μπέιζιγγεν και στην Χάλε, στο Βέλιο, που προκάλεσε το θάνατο πολλών ατόμων, μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Ήταν ένα μέλος του προσωπικού του Κοινοβουλίου, ο Κλάουδιο Καντιέγο, ...40 ετών, στην ομάδα τύπου και μέσων ενημέρωσης, στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Η τραγική αυτή λοιπόν συνδρομική σύγκρουση ήταν τραγική και για το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να κρατήσετε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη αυτών που χάσαν τη ζωή τους. Φυσιολογικά θα πήγαμε στην ημέρησια διάταξη κατευθείαν. Ξέρω ότι κάποιοι από του Βέλγου συναδελφού μα θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια. Συμφώνησα λοιπόν προ ημερήσια διάταξη να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο. Κύριο Στάς θα ήθελα να λάβει το λόγο από ό,τι βλέπω. Ντέρκ, θες να ξεκινήσει και μετά ο Σαΐντ να συνεχίσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που επιτρέψατε στην Επιτροπή μας να αποτίσει φόρο τιμής στους θανόντες. Η κατάσταση είναι βέβαια δραματική. Η ακριβή αιτία του ατυχήματος δεν είναι απόλυτα γνωστή, συνεχίζονται οι έρευνες. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η γραμμή η σειροδρομική είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε σύγκριση με άλλες και μια τέτοια καταστροφή είναι φοβερή. Οι αρχές της χώρας μου θα φροντίσουν, δίχως άλλο, να ξεκαθαριστούν τα αίτια του ατυχήματος και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια στις δρομικές γραμμές. Τώρα, η συζήτηση βέβαια πρέπει να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των συνδρομικών γραμμών. Για μένα, έχοντας μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ε, που ξέρουν ε, από τα πράγματα, έχουμε ακούσει διάφορες παρατηρήσεις. Η δικιά μου παρατήρηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αλήθεια ότι δεν έδωσε σημασία στην ασφάλεια. Εγώ ο ίδιο ήμουν εισηγητή εδώ σε αυτή την επιτροπή όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και εκεί είχαμε υπογραμμίσει την ασφάλεια και ότι έπρεπε να έχουμε τις υψηλότερες δυνατόν προδιαγραφές. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή που σε συνεργασία με το Συμβούλιο φροντίζει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η συζήτηση συνεχίζεται βέβαια. Τα συλληπιτήριά μου εννοείται όχι μόνο για τις οικογένειες των ε, θανόντων, αλλά και ε, θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες που είναι ακόμα πολλοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Στέρκ. Πρέπει να πω ότι εγώ ε, απογοητεύτηκα πάρα πολύ όταν ακούστηκαν διάφορες υπόνοιες μετά το ατύχημα από διάφορες οργανώσεις στο Βέλιο που μίλησαν σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι φταίει δηλαδή. Οπότε συμφωνώ με αυτά που είπατε σήμερα. Ας αρκεστούμε σε αυτό. Σαΐτ, ευχαριστώ. Ναι, είναι και η σειρά μου τώρα και εγώ εκ μέρους της ομάδας μου θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου όσον αφορά τα θύματα του ατυχήματος αυτού. Όπως είπε και ο συνάδελφος Dirk Sterks, είναι ασφαλεί οι σιδηρόδρομοι, αλλά βέβαια όταν συμβεί κάποιο ατύχημα οι συνέπειε είναι τεράστιες. Δικός μας ρόλος λοιπόν εδώ είναι να συζητήσουμε για το ποιο είναι υπεύθυνο, για το τι θα έπρεπε να γίνει, τι έφτεξε και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο εμείς να αποφανθούμε από αυτού. Πάντως η Επιτροπή μας πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Έχουμε ήδη κάνει πολλά, αλλά είναι ένα, μια δουλειά που θα κρατήσει πολύ. Πρέπει να δούμε τι σύστημα πρέπει να εφαρμόσουμε. Είναι κάτι που συζητιέται στο Βέλγιο αυτή τη βδομάδα, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να διασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Σίγουρα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας σε τι βαθμό οι ευρωπαϊκές σιδηροδρογραμμές μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς και καλύτερες για όλους μέσα στην Ευρώπη. Να το συζητήσουμε λοιπόν, φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Ντουρά, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω πολλά από αυτά. Πέραν αυτών που είπαν οι συναδελφοί μου, είναι γεγονό ότι τόσο από σεβασμό για τι οικογένειε των θανόντων και για το κοινοβούλιο που έζησε και αυτό το τμήμα αυτό τη καταστροφή, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την διαλεύκανση του θέματος αυτού. Εγώ ενοχλήθηκα από το γεγονός ότι οι άλλοι δακτυλοδεικτούσαν το Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι το Βέλγιο ως υπευθύνους. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες να βελτιωθεί η συνδεδομική ασφάλεια για να υπάρξει και μεγαλύτερη εναρμόνιση, για να υπάρξει καλύτερη υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη και τις συνδρομικές εταιρείε για να λειτουργήσουν καλύτερα συστήματα ασφαλιών θα πρέπει να σκεφτούμε και τις συνθήκες εργασίας των μηχανοδηγών. Αυτά είναι θέματα που αφορούν όχι μόνο το Βέλγιο, αλλά και άλλες χώρες. Ευτυχώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τους σιδηροδρόμους. Αυτό όμως σημαίνει και μεγαλύτερη πίεση στους μηχανοδηγούς και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων αυτών και όλων των ε, μεταφερομένων με σιδηρόδρομο, αν θέλουμε λοιπόν να είναι ευχάριστη η σιδηροδρομική μεταφορά και αποτελεσματική. Αυτός είναι ο στόχος που όλοι μας θέλουμε να υποστηρίξουμε στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε όλες τις πτυχές της συνδρομικής ασφάλειας και σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο χρόνου εργασίας και συνδικών εργασίας των μηχανοδηγών. μετά από τους Βέλγους συναδέλφους, ήταν και άλλοι συναδελφοί που ήθελαν να λάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι, καταλαβαίνω το πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό αλλά θα ήμουν ευγνώμων αν μπορείτε να είσαστε σύντομοι. Ο κύριος Στούσας και ο κύριος Κούν. Θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και θεωρούμε ότι καλύτερη τιμή στη μνήμη αυτών που έχασαν τη ζωή τους είναι να σχεδιάσει, να προγραμματίσει η Επιτροπή μας μια ολοκληρωμένη συζήτηση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και διαπιστώνεται αύξηση των ατυχημάτων. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε σκέψεις αλλά και να προτείνουμε μέτρα. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω κύριε Τούσα, ευχαριστώντας σας, ότι είχαμε επανειλημμένα συζητήσει επί του θέματος αυτού στην Επιτροπή μας, ο κύριος Κούν. Εξ του ΕΛΚ και εγώ θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής και να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς οικογένειες των θανόντων και των οικείων τους Και ιδίω θέλω να τονίσω ότι πολλοί από εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσω μόνο από καλή τύχη γλιτώσαμε. Θα μπορούσαμε και εμεί να ήμασταν, οι γνωστοί μα και οι φίλοι μα να ήταν μέσα σε αυτό το ατύχημα. Όπω έχουμε κάνει λοιπόν πολλέ φορέ στο παρελθόν, θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι η ασφάλεια στο, στις συνδρομικές μεταφορές και ιδίως στις ε, συνδρομικές γραμμές οι οποίες είναι κοντά στην πρωτεύουσα των Βρυξελών θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και εμεί θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στου οικείου του μέλου του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στι οικογένειε όλων των θυμάτων. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε για τον τρόπο που αντιμετώπισε το θέμα, αντιμετώπισαν τα βελικά μέσα ενημέρωση σε αυτό το θέμα αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να αντλήσουμε τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικών ή δεν είναι το θέμα των δημοσιογράφων. Χρειάζεται γαλήνη, χρειάζεται προβληματισμός και όχι να προσπαθούμε να έχουμε πηχαίους τίτλους και δημιουργία εντυπώσεων. Κάτι που μπορείτε να κάνετε λοιπόν ως πρόεδρος της Επιτροπής μας είναι να αποστείλετε μια επιστολή εξ ονομότητας της Επιτροπής μας στις αρμόδιες βελγικές αρχές για να τονίσετε την άποψή μας ότι πιστεύουμε ότι χρειάζεται γαλήνη και υπομονή ώστε να μπορέσουν οι απαραίτητες, οι αντίστοιχες αρχές να καταλάβουν τι συνέβη για να αποτραπεί και στο μέλλον η επανάληψη αυτού του φαινομένου θα είναι η πρόθεσή μου με την έγκρισή σας βέβαια να γράψω στο Βελικό Υπουργείο Μεταφορών να εκφράσω την, τα συλληπιτήριά μας για αυτό το τρομερό συμβάν και επίσης να εκφράσω την θέλησή μας να αναμείνουμε την επίσημη την έκθεση για το γεγονός αυτό προτού καταλήξουμε σε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Κάθε φορά που γίνεται ένα ατύχημα προτρέχουν όλοι και προσπαθούν να βρούνε μια εξήγηση. Θα ήταν χρήσιμο όμως να περιμένουμε περισσότερο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Κατανοώ πάντως τις απόψεις και είναι σαφές ότι η Επιτροπή μας έχει κάθε συμπάσχει πλήρως με όλους αυτούς οι οποίοι ήταν οι επιβάτες, η σιδηροδρομικό προσωπικό που έχασαν τη ζωή τους και ελπίζουμε ότι οι βελικές αρχές θα καταλήξουν σύντομα σε συμπεράσματα για τα αίτια του ατυχήματος αυτού. Σας ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο, στην ίδια την ημερησία διάταξη. Από ό,τι γνωρίζω, χαθήκανε κάποια τα φορτηγά μας μεταξύ Λουξεμβούργου και Βρυξελών και δεν έχουμε αρκετούς φακέλους. Ο κύριος Φαντάλεν θα λάβει το λόγο στη συνέχεια, αλλά οι φάκελοι μας κάπου έχουν ξεμείνει μεταξύ Λουξεμβούργου και Βρυξελών. Που κυρία Φώστερ δείχνει ότι δεν είναι μονάχα η Αγγλία η οποία παραλύει όταν χιονίζει, αλλά και άλλες χώρες. Το ταχύτερο δυνατό λοιπόν μόλις φτάσουν οι φάκελοι θα σας τους διανύμουμε. Ερχόμαστε λοιπόν στην έγκριση της ημέρησης διάταξης. Δεν έχει αναφέρει κανείς ότι θέλει να κάνει κάποια τροποποίηση. Νομίζω ότι αν συμφωνείτε μπορούμε να αποδεχθούμε την ημερησία διάταξη. Τα πρακτικά της 25ης με 27η Ιανουαρίου. Εάν δεν έχετε αντίρρηση και εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε στο θέμα του κύριου Φαντάλεν για την θαλάσσια πολιτική. Συγγνώμη κύριε Φαντάλεν που καθυστερήσαμε λιγάκι, ξέρετε γιατί αλλά έχετε τώρα πλέον το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου σήμερα, εδώ. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δούλεψα με πολύ χαρά το θέμα αυτό, έτσι και με το χαμηλό φωτισμό, Ξεκίνησα λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά, λέω, να δουλεύω αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία να πάρω έγγραφα, να τα μελετήσω. Είναι καλό που έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να εξετάσουμε αυτό το θέμα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η οποία δεν έχει τελειώσει. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας δύσκολης χρονιάς, αλλά και συγχρόνως οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Το ξέρουμε αυτό από τους τελευταίους μήνες. Πολύ σημαντικό αυτό και για την ασφάλεια στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό μέσα στα επόμενα χρόνια να δούμε τι είναι σημαντικό όσον αφορά την ασφάλεια στις θάλασσές μας, την ασφάλεια των πλοίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές. Είχα την τιμή λοιπόν να είμαι και να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε γρήγορα και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις. Έρχομαι στο κύριο θέμα, που, στο οποίο θέλω να πιστήσω την προσοχή σας. Και θα τα βρείτε όλα αυτά βέβαια στην έκθεσή μου. Θα υπογραμμίσω μερικά σημεία μόνο. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τομέας αυτός έχει μια παγκόσμια διάσταση. Συζητάμε για διάφορα είδη μεταφορών στην Επιτροπή μας, θαλάσσιες, αλλά και για τα ποταμόπλια, στα εσωτερικά ύδατα, για την αεροπορία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα παγκόσμιο είδος μεταφορών που πλήττεται από το παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και αυτό το εξηγώ στην έκθεσή μου. Ξεκινάω λοιπόν με αυτό και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, την παγκόσμια διάσταση του θέματος. Το δεύτερο είναι πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ίδιος ο τομέας. Είναι ζωτικής σημασίας να το υπογραμμίζουμε στην έκθεση ότι η θαλάσσια ναυσιπλοεία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για την καθημερινή ζωή του καθενός μας. Διότι μεταφέρονται αγαθά, επιβάτες, με τις θαλάσσιες μεταφορές. Πράγματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ποτέ δεν το υπογραμμίζουμε αρκετά αυτό. Τρίτον, κάτι άλλο που αναφέρω στην έκθεση είναι το θέμα των κρατικών ε, επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων. Με την Επίτροπο το θέμα αυτό το συζητάμε. Αλλά παραμένει ένα θέμα κλειδί όταν πρόκειται για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τον τρόπο με τον οποίο δίνονται ή μπορούν να δίνονται οι κρατικές ε, επιχορηγήσεις. Τα αναφέρω αυτά στο σχέδιο εκθεσής μου. Ο Επίτροπος Κάλλας έκανε πολλά μέχρι τώρα, αλλά τους επόμενους μήνες μένουν να γίνουν πολλά ακόμα. Βέβαια σε συνεργασία με τη, τον συνάδελφο για τον ανταγωνισμό πρέπει να δουλευτεί ακόμα αυτό το θέμα για να εξεταστούν όλες οι πτυχές των κρατικών επιχορηγήσεων. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι αυτή για την οποία κάνω προτάσεις και θεωρώ πολύ σημαντική να προσέξουμε. Στην Ευρώπη έχουμε ένα δημογραφικό ζήτημα. Ο πληθυσμός μεγαλώνει σε ηλικία και αυτό πρέπει να μας κάνει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες εργασίας στα πλοία. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για τα πλοία, πρόκειται και για ένα σώρο επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, βρίσκονται δίπλα από την έρευνα μέχρι άλλα επαγγέλματα στη θάλασσα. Και έτσι όλα αυτά μαζί πρέπει να τα εξετάσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, να μην τα ξεχνάμε. Μην μιλάμε δηλαδή μόνο για τις μεταφορές. Ένα άλλο σημείο που με ενδιαφέρει εδώ είναι ο έλεγχος. Τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις να εξακολουθούν να γίνονται, να μην μειωθεί, να μην πέσει η ποιότητα, αλλά από την άλλη μεριά οι απαιτήσει από τους ελέγχους να μην είναι τέτοιοι που να πλήττουν τον ανταγωνισμό. Πρέπει λοιπόν ίσω να βρούμε μια νέα μεθοδολογία για να εξετάζουμε τον κίνδυνο και να εκτιμάμε τον κίνδυνο. Έχω συζητήσει με διάφορου συναδέλφου που βρίσκουν ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά και εγώ ίδιο, στο θέμα του περιβάλλοντο. Σίγουρα, όταν πρόκειται για μεγάλα πλοία και για διπυρωτικέ μεταφορέ, Από την άλλη μεριά υπάρχει και η εκτοπλοεία με μικρότερα σκάφη που είναι πιο σύγχρονα με σύγχρονους κινητήρες που δεν προκαλούν ιδιαίτερη ζημιά στο περιβάλλον. Πάντως θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πρέπει να αναπτυχθεί νέα τεχνολογία. Έχω κοιτάξει λίγο τι ισχύει στις μεταφορές της θαλάσσιας, όχι μόνο μάλλον στη θάλασσα, αλλά και στα εσωτερικά ύδατα και υπάρχουν νέοι κινητήρε, τουλάχιστον ε, που έχουν τα ποταμόπλια και που ίσως θα μπορέσει αυτή η τεχνολογία να αναπτυχθεί περισσότερο για να εφαρμοστεί και στη θάλασσα. Να έχουμε τέτοιου κινητήρες δηλαδή και στα σκάφη της ε, θάλασσας. Έπειτα υπάρχει και η έννοια των πράσινων λιμένων όπου ίσως θα μπορούσαν τα καθαρά σκάφη, αυτά τα οποία δεν προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον, να πληρώνουν λιγότερα χρήματα για να μπαίνουν στους λεγόμενους πράσινους λιμένες. Να βρούμε κάποια τέτοια μέτρα υπέρ των καθαρών σκαφών. Είμαι έτοιμος να ακούσω προτάσεις από τους συναδέρφους, συστάσεις και τέλος όσον αφορά τον οδικό χάρτη, η Επιτροπή έχει κάνει την πρότασή της. Εγώ θα ήθελα να ξέρω περισσότερα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Τέλος, θα ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ό,τι σχόλια και προτάσεις έχουν να κάνουν οι συνάδελφοι για τη δικιά μου την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βανάμ. Ε, μία παράκληση, αν μπορούμε να, μιλήσουμε, να χαμηλώσουμε λίγο τη θέρμανση. Ε, συνήθως μου λέτε ότι είμαι κρύος και ψύχρεμος, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, παρότι έχω κρύο αίμα, τώρα θα ήθελα λίγο να χαμηλώσουμε τη θέρμανση. Ε, λοιπόν, από το ΕΛΚ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που ξεκινάει στην Επιτροπή μας και ευρύτερα στο Κοινοβούλιο με την ε, αφορμή της πρότασης του ψηφίσματος για τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσει πολιτικής για μια ευρωπαϊκή πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018 είναι εξαιρετικά σημαντική. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία που ε, διέρχεται η διεθνής οικονομία και οπωσδήποτε επηρεάζει την ευρωπαϊκή ναυτιλία θα συμφωνήσω με τις βασικές παραδοχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της ε, τοποθέτησης αλλά και του σχεδίου που έχει παρουσιάσει ο κύριος ε, Βαντάρλεν. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένες επισημάνσεις και ορισμένα σημεία που χρειάζονται ενδεχομένως λίγη περισσότερη <clears throat> συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις συν μία προκλήσεις. Οι τρεις αφορούν την ίδια την ναυτιλία και η μία αφορά, αν θέλετε, είναι ένας εξωγενής παράγοντας. Οι τρεις προκλήσεις είναι πρώτα απ' όλα η ανάγκη βελτίωσης του έμψυχου δυναμικού των εργαζομένων στην ναυτιλία. Και η βελτίωση της ποιότητας, αλλά και οπωσδήποτε η μεγαλύτερη προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα νέων επαγγελματιών σε αυτόν τον τομέα είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, διότι οι αριθμοί δυστυχώς δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μια μείωση ενδιαφέροντος στους νέους Ευρωπαίους για να εργαστούν σε αυτό τον πολύ κρίσιμο για την ευρωπαϊκή οικονομία τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι για να αντιστραφεί ή εν πάση περιπτώσει σε πρώτο στάδιο να συγκρατηθεί αυτή η κατάσταση μεταξύ των σκέψεων που κανείς θα μπορούσε να κάνει είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένα, ε, να καταρτιστούν ορισμένα προγράμματα μακροπρόθεσμα για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων επί των πλοίων. Παραδείγματος χάρη θα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών των πληρωμάτων ώστε να βληθούν τα προβλήματα αλλά και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κόπωση. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε εάν μπορούμε με κάποιο τρόπο να καθορίσουμε τον ελάχιστο αριθμό των μελών του πληρώματος. Αυτά τα αναφέρω μόνο ως ενδεικτικά στοιχεία μιας ευρύτερης πολιτικής που πρέπει να γίνει για την προσέλκυση ε, περισσότερων <clears throat> στο επάγγελμα του ναυτικού. Τώρα, η δεύτερη πρόκληση είναι βεβαίως ο διεθνής ανταγωνισμός και εκεί πρέπει να πούμε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία, επειδή έχει θέσει πολύ υψηλά standards, πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αθέμητο ανταγωνισμό, πράγμα το οποίο βαίνει εις βάρος της, ενώ από τρίτες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τι θα γίνει με το θέμα των, ε, πιθανών ενισχύσεων στο μέλλον. Ξέρω ότι ο κύριος, ο στο report του είναι επιφυλακτικός γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει σοβαρά να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ενισχυθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ή ε, ε, ναυτιλία. Και ίσως σε αυτή την έκθεση και επειδή ο ορίζοντας είναι το 2018 θα μπορούσαμε υποτύπων προτροπής να καταγράψουμε ότι αυτές οι ενισχύσεις στο μέλλον θα πρέπει καταρχήν να χορηγούνται σε πλοία που φέρουν σημαίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρίτη πρόκληση είναι βεβαίως τα θέματα περιβάλλοντος και πώς η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές ε, επιβαρύνουν με το δικό τους ποσοστό ε, τα θέματα το, το περιβάλλον. Εδώ πρέπει να πω ότι η έκθεση του κυρίου Βαντάλεν περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Είναι αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 16 ένα είδος μπόνους μάλους για τα ε, πλοία τα οποία είναι πιο φιλικά ε, στο περιβάλλον. Η πρόταση παρόλα αυτά νομίζω ε, ότι παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει θα πρέπει να συζητηθεί και να μας απασχολήσει λίγο περισσότερο. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε το χρόνο στο πλαίσιο της ζήτησης που θα κάνουμε στην Επιτροπή να, να δούμε και να μας πει και ο κύριος Βαντάλεν πώς βλέπει περισσότερο και πιο συγκεκριμένα τη συγκεκριμένη του πρόταση. Επίσης, ίσως θα χρειαστεί μία διευκρίνηση ε, του στοιχείου που αναφέρεται στο πρώτο τμήμα της παραγράφου 16, που, στην οποία καλείται η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν άλλα μέσα, όπως η εισαγωγή ενός φόρου επί των καυσίμων στη δεξαμενή, κατά προτίμηση υπολογιζόμενο στη βάση ποιότητα και περιβαλλοντολογική σημαντότητα των καυσίμων. Είναι λιγάκι ασαφής αυτή η ιδέα. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Βαντάλεν θα μπορούσε να την εξειδικεύσει και θα πρέπει να δούμε λιγάκι περισσότερο ε, πώς ακριβώς εννοείται αυτό. Ε, κατά τα λοιπά, όσον αφορά το περιβάλλον, συμφωνώ με τη γενική φιλοσοφία του κειμένου του κ. Βαντάλεν, και άφησα, αυτή ήταν η τρίτη πρόκληση αν θέλετε που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία, άφησα για το τέλος αυτό που ανέφερα στην αρχή ως τρεις προκλήσεις συν μία. Η η μία αυτή πρόκληση που είναι περισσότερο εξωγενής, δεν ανήκει μέσα στον τομέα της ναυτιλίας, είναι η διεθνής πειρατεία. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκω όχι τόσο φιλόδοξη την έκθεση του κ. Βαντάλλα όταν αναφέρεται στην καταπολέμηση της διεθνούς πειρατεία στη θάλασσα. Η παράγραφος 25 η οποία αφιερώνεται στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου ε, μου φαίνεται ότι επιδέχεται μεγαλύτερης ανάπτυξης και μπορεί να εμπλουτιστεί με περισσότερες ιδέες και κατευθυντήριες γραμμές. Εδώ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην στενή αρμοδιότητα της Επιτροπής, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ή να συζητήσουμε ιδέες όπως μεγαλύτερη συνεννόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του φαινομένου, καθώς επίσης ε, να εντάξουμε σκέψεις όπως η ανάπτυξη της αναπτυξιακής βοήθειας και ε, τελειώνω προς τις χώρες από τις οποίες πηγάζει κυρίως το φαινόμενο της ναυτιλίας. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει για την, ε, της τι σημαίνει για την πειρατεία και την καταπολέμησή της η έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας και αρμόδιων δικαστηρίων που μπορούν να δικάσουν θέματα, το φαινόμενο της πειρατείας και όσων εμπλέκονται σε αυτήν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ήταν μια συνολική ε, πρώτη προσέγγιση του πολύ ενδιαφέροντος κειμένου που έχει παρουσιάσει ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Φαντάλεν για την πλήρη αυτή έκθεση που μας παρουσίασε Έχουμε λοιπόν μια εκτενή και εμπεριστατωμένη έκθεση για τα ζητήματα αυτά. Και θα θέλαμε βέβαια να έχουμε το ταχύτερο δυνατόν και το νομοθετικό σχέδιο δράσης της Κομισιόν, τον οδικό χάρτη της Κομισιόν για την έκδοση νομοθετημάτων στο θέμα αυτό. Και φυσικά τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μια επίπτωση στη Λευκή Βίβλο της Κομισιόν για τα θέματα της, ε, της ναυτιλίας. Σίγουρα υπάρχουν σημεία στα οποία συμφωνούμε όλοι, δεν θέλουμε να ευνοηθεί η αλλαγή σημαία, θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πλοίων. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να κάνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και όχι απλώς να συζητάτε μόνο προτάσεις, αλλά να τις εφαρμόζει και στην πράξη. Επίσης, ό,τι αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις, μπορούμε να σταθούμε σε πιο πολύ λεπτομέρεια για τους τομείς στους οποίους εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, ώστε να υπάρξουν ε, να υπάρξει μια ειδική αντιμετώπιση για τα πλοία τα οποία φέρουν ευρωπαϊκή σημαία. Και ο στόχος μας είναι οι κατευθυντήρες γραμμές για όλα αυτά τα θέματα να μας ανακοινωθούν από την Κομισιόν μέχρι τον Αύγουστο του 2010 όπως έχει αναφερθεί, ώστε να υπάρχει και μία σαφήνεια σε σχέση με τις προτινόμενες επιχορηγήσεις για τους θαλάσσιους λιμένες. Εγώ λοιπόν θα μπορώ να είμαι σύντομο γιατί σε κάποιο βαθμό επαναλαμβάνω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντε για τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αναφερθήκαμε καταρχήν στο θέμα τη κατάρτιση σε ό,τι αφορά το προσωπικό των ε, θαλασσίων μεταφορών. Εδώ θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις απλές δηλώσεις προθέσεων και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε από την Κομισιόν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράση το οποίο θα θεραπεύσει αυτή την έλλειψη ναυτικών. Δεύτερον, για το περιβάλλον θέλουμε φυσικά εμείς να περιλάβουμε και την ε, ναυτιλία στον χώρο παρακολούθησης των εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές. Αλλά όταν το πράξουμε αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε πάντα δύο πράγματα στο μυαλό μας. δεν θέλουμε να αυξήσουμε τόσο πολύ το κόστος θαλασσίων μεταφορών που να πάψει να είναι πια ε, ελκυστική η ναυτιλία ως μέσο μεταφοράς και να φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν κάποιες τις θαλάσσιες μεταφορές από οδικές μεταφορές και επίσης θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να μπορεί η ευρωπαϊκή ναυτιλία να είναι ανταγωνιστική, να διατηρηθεί μια ισότης ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις βραχίες τώρα θαλάσσιες μεταφορές, χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή εκμετάλλευση του δυναμικού για βραχίες θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως όμως αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο το θέμα αυτό. Και επίσης σε ό,τι αφορά την ε, πτυχή και του περιβάλλοντος και πάλι στην οποία επανέρχομαι. Έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα μέτρα για την ε, μείωση της επίπτωσης των πλοίων στο περιβάλλον, αλλά δεν έχουμε ακόμα τέτοια, τέτοια μέτρα. Πάντως χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη στρατηγική για τι θαλάσσιες μεταφορές μεταφορέ και επίσης για την μεταφορά με εσωτερικέ θαλάσσιες οδού. Ένα τελευταίο σημείο. Θα πρέπει να σκεφτούμε και για την εντολή της ΕΜΖΑ. Η ΕΜΖΑ θα πρέπει να έχει σαν στόχο την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών στις θαλάσσιες μεταφορές. Έχουμε τη δυνατότητα η ΕΜΖΑ να είναι ενεργή και στον τομέα του περιβάλλοντος, μια ευκαιρία που δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Θα πρέπει όμως για να επιτευχθεί αυτό να υπάρχουν και ευρύτερες αρμοδιότητες της ΕΜΖΑ. Παράδειγμα, η ΕΜΖΑ ελέγχει μεν τα, τις σχολές για, τις, για τους αξιωματικούς στα πλοία, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάρτισης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι λογικό να περιορίσουμε τη δυνατότητα της ΕΜΖΑ να επηρεάζει τα θέματα κατάρτισης. Και ένα τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να, θέσω η συμπερίληψη της ναυτιλίας στα διευρωπαϊκά δίκτυα και το σχεδιασμό των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να ενισχυθεί γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητη για να υπάρχει μια σωστή σχεδιοποίηση που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς θαλάσσιες μεταφορές. Ναι, φαίνεται ότι φτάσανε τα φορτηγά. Έχουμε και τα χαρτιά μας. Ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάβη Σαρίνης και η συγκήτριά μας, αλλά δεν είναι εδώ μάλλον έχει πρόβλημα με τις μεταφορές. Οπότε εγώ θέλω να πω στον κύριο Βαντάλεν ότι συμφωνούμε με την εκθεσή του, η ομάδα μας δηλαδή. Και χαίρομαι που υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι θαλάσσιες μεταφορές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από την οικονομική άποψη, αλλά και όσον αφορά την καινοτομία. Και είναι σημαντικό, λοιπόν, να δούμε την προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Και είναι καλό να υπάρχουν και τα δύο, να υπογραμμίζονται και τα δύο. Και κυρίω χαίρομαι που ο εισηγητή δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό στοιχείο για την όλη εξέλιξη του τομέα. Η ποιότητα του σκάφους εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό και από το πλήρωμά του. Και χαίρομαι που έχει αυτή την προσέγγιση στο κείμενό του εισηγητή. Ευχαριστούμε, κύριο Πεσέ. Δύο παρατηρήσεις μονάχα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Συγητά. Δύο παρατηρήσεις λοιπόν σύντομες, διότι η έκθεσή σας ε, θίγει πολλά ενδιαφέροντα και θετικά στοιχεία. Θα θέλαμε η έκθεση αυτή να προσανατολιστεί περισσότερο προς την ιδέα της ευρωπαϊκής θάλασσας, δηλαδή ενός ευρωπαϊκού ε, θαλασσίου χώρου και επομένως ε, οι στόχοι ε, για το 2018 όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές να ε, ειδωθούν ακριβώς σε σχέση με αυτόν τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο. Δεύτερη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το ζήτημα το, της μείωσης των ε, εκπομπών κυρίως αζότου και οξυδίου ε, του θείου. υπογραμμίζεται λοιπόν στην έκθεσή σας και συγκεκριμένα στο σημείο 14 ότι αυτά τα μέτρα μείωσης τα οποία συμμεριζόμαστε θα πρέπει να εγκριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι ε, πιστεύετε ότι αυτές οι μειώσεις θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο πριν τις εφαρμόσουν ε, τα ε, πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εμείς φρονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα και να μπει μπροστά στον αγώνα για την καταπολέμηση της μόλυνσης. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Μερικά πολύ σύντομα σημεία. Ε, θεωρούμε ότι ο κύριος Βαντάλεν έκανε εξαιρετικά καλή δουλειά όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης του. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια ε, σημεία από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίως συμμεριζόμαστε ε, τα μελήματα της, και τις Ανησυχίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Επιτροπής μας εδώ όσον αφορά τα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά ακριβώς την παγκόσμια ναυτιλία. Επίσης, οτιδήποτε ε, αναφέρεται σε ε, προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή ε, Οργανισμό Ναυσιπλοείας θα πρέπει να ειδωθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αντιθέτως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το IMO έτσι ώστε να προωθήσουμε καλύτερα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί καλύτερα η αναφορά ε, στις επαφές που θα πρέπει να έχουμε με τα ενδιαφερόμενα ε, μέρη και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εκείνοι να επικυρώσουν οι συμφωνίες. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι ε, όσον αφορά το θέμα των σημεών νομίζουμε ότι δεν υπάρχει λόγος, αλλά δεν έχουμε και μεγάλο πρόβλημα να δούμε και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις άλλες σημείες. Ο κύριος Τούσας. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι και συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές» καθορίζει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο στόχος της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου, συνολικά του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον ναυτιλιακό τομέα και στους συναφείς κλάδους. Γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση και στην έκθεση του εισηγητή σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Δεν γίνεται όμως καμία αναφορά τόσο από την εισήγηση της Επιτροπής όσο και από την έκθεση του εισηγητή σε ό,τι αφορά ότι το 80% των, της πλειοκτησίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά βρίσκονται σε σημεία της ευκαιρίας. Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ε, Γερμανία, Ολλανδία. Αλήθεια, ποιος μπορεί να αποσιωπήσει τέτοια σοβαρά στοιχεία που καταγράφονται και αναγνωρίζονται από διεθνείς οργανισμούς. Όσο και από τη μελέτη που επικαλείται για να τεκμηριώσει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής όσο και ο εισηγητής. Εδώ πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για εμπεγμό. Δηλαδή οι εφοπλιστές ανταγωνίζονται την αριστερή με τη δεξιά τους τσέπη. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Από ό,τι έχω υπόψη μου έχει γίνει συζήτηση στο επίπεδο της ΣΟΚΕ για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος χρειάζεται να παρθεί σοβαρά υπόψη γιατί αυτές οι ναυτιλιακές εταιρείε εκμεταλλεύονται τις υποδομές, εκμεταλλεύονται τις ανάγκες ε, της εισαγωγής πρώτων υλών, της εξαγωγής εμπορευμάτων, όλες τις διαδικασίες που πραγματικά απασχολούνται και αποκομίζουν τεράστια κέρδη πέρασαν μια μεγάλη φάση και περίοδο Σεπτέμβρης 2003, Ιούλης 2008 με αστρονομικά κέρδη. Μάης του 2008 Cape Size πλοίο 204.000 δολάρια ημερήσεως ναύρος των πλοίων. Το πρώτο στοιχείο που επικεντρώνεται η εισήγηση της Επιτροπής και του εισηγητή είναι σε ό,τι αφορά τον αφεργατικό δυναμικό και δείχνει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την έλλειψη αξιωματικών στα πλοία. Αφού τα προηγούμενα χρόνια τους αντικατάστησαν, τώρα πραγματικά φαίνεται η έλλειψη και οι επιπτώσεις που έχει αυτή. Αν και σε ό,τι αφορά τα κατώτερα πληρώματα έχουν εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό, πλέον δεν τους ενδιαφέρει, αφού μπορούν να τα αντικαταστήσουν με πιο φτηνότερο εργατικό δυναμικό 550 δολάρια το μήνα ο ναύτης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 του IMO. Μπαίνουν σοβαρά ζητήματα. Μπορώ να σταματήσω. Αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει χρησιμότητα να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Μπαίνουν ορισμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Μπαίνει εδώ το ζήτημα της αξιοποίησης της πράσινης οικονομίας και στον τομέα της ναυτιλίας. Μπαίνουν και εδώ ζητήματα που θα πρέπει να δοθούν ε, επιδοτήσεις στους εφοπιστές ε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία πλοίων που πραγματικά θα ε, αξιοποιούν και θα χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία. Το θέμα είναι το εξής. Για να έχει αποτέλεσμα η συνολική ναυτιλιακή πολιτική σε ό,τι αφορά την προστασία του, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να επιμείνουμε σε ό,τι αφορά να παρθούν μέτρα στο επίπεδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ε, είναι ένα ζήτημα πολύ ανοιχτό που πραγματικά ο δικός χάρτης που θα προταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα προφανώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, την αφιλία πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά και με την οργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε ολοκληρωμένα να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με αυτό κύριε Πρόεδρε κατανοώ και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε αλλά να τελειώσω με το εξής. Τι θα γίνει με τις αρτοπορικές συγκοινωνίες. 370% μέσα σε πέντε χρόνια αύξηση της τιμή των εισιτηρίων. Δεκαπλασιασμός των επιδοτήσεων των επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στην ξέρα. Ποιοι είναι αυτοί που καρπώνονται όλο αυτό το πλούτο. Άρα λοιπόν προκύπτει από όλη αυτή την πρώτη συζήτηση ότι χρειάζεται πιο διεξοδικά να συζητήσουμε και να πάρουμε μέτρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βαν Τάλεν για την έκθεσή του και θα ήθελα να κάνω και ορισμένα σχόλια. Σε ό,τι αφορά καταρχήν την ε, πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία των διαφορών φορέων που εμπλέκονται στις μεταφορές. Όχι μονάχα να υπάρξει λοιπόν συνεργασία σε επίπεδο θαλασσίων λιμένων, αλλά και των θαλασσίων λιμένων με τους ποτάμιους λιμένες που είναι σε εκβολές ποταμών. Επίση, η έκθεση του κ. Φαντάλεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα θέματα βιομηχανική πολιτική και αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου είναι η βιομηχανική πολιτική η οποία συνδέεται με την πολιτική των θαλασσίων μεταφορών. Παραδείγματο χάρη τα ναυπηγεία. Δεν είναι μονάχα θέμα θέσεων εργασία και του να υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό, αλλά και σε ό,τι αφορά την πρόθεση της παραγωγής. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραστικά η ναυπηγική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημείο επίση, το οποίο ανέφερε ο κύριος ε, Φαντάλεν και το οποίο έχει να κάνει και με την οικονομική ανάπτυξη. Η, το θέμα των ελευθέρων, των λεγόμενων ελευθέρων λιμένων. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει και κάποια μνήμα αυτών των λεγόμενων ελευθέρων λιμένων στην έκθεση του κυρίου Φαν και επίσης να αντιμετωπιστούν τα θέματα της ασφαλείας της θαλάσσιας μεταφορές. Χρειαζόμαστε να έχουμε και κέντρα ταχείας επέμβασης σε περίπτωση ατυχημάτων. Θα μπορούσαμε στην περίπτωση του εύξηνου πόντου να έχουμε ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Κάτι το οποίο επίσης συνδέεται με το θέμα της ασφάλειας είναι και η καταπολέμηση της πειρατείας. Υπάρχουν όμως κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία βρίσκονται στην μαύρη λίστα ή στην γκρίζα λίστα του Μνημονίου των Παρισίων για τη θαλάσσια ασφάλεια. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να βελτιωθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε ό,τι αφορά την τήρηση των προτύπων και να μπουν οι χώρες μας όλες στη λευκή λίστα. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι υπάρχουν όπως ελέγχθη κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στον γκρίζο και το μαύρο κατάλογο του ΙΜΟ. Αυτό εντάξει, το κατανοήσαμε κυρία Τικάου ο κ. Θεολογάκης από την Κομισιόν. Τα ελληνικά μου προσπαθώ να τα βελτιώσω γιατί ξέρω ότι έχει πολλά ελληνικά ονόματα. Θεολογή της κύριε Πρόεδρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πολύ καλή προσπάθειά σας και με κολακεύετε. Από την πλευρά της Κομισιόν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή τον κύριο Νταφάν Ντάλεν για τα θετικά σχόλιά τους σε σχέση με το έργο της Επιτροπής. Η ανακοίνωση της Κομισιόν είναι το αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης και με τους εργαζόμενους του τομέα και τις επιχειρήσεις και με τις δημόσιες αρχές, με στόχο να αντιμετωπίσει τα θέματα που έχουν θίξει όλοι οι συνομιλητές μας. Και νομίζω τα σχόλια του κ. Φαντάλεν καταδεικνύουν και την προσπάθεια και την φροντίδα που έχει μπει στην έκθεση αυτή από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν πρόκειται τώρα να διεξέλθω όλα τα σημεία τα οποία ανέφεραν οι ομιλητές. Μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η Κομισιόν βρίσκεται ήδη εν μέσω εργασιών για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά που ανέφεραν όπως το να γίνει ελκυστικό το επάγγελμα του ναυτικού, η περαιτέρω ανάπτυξη της ασφάλειας πλοήγησης, η καταπολέμηση της πειρατείας, τα θέματα της ε, ανταγωνιστικότητες που έχουν να κάνουν με το φορολογικό καθεστώς για την αυτιλία που τώρα σιγά σιγά μπορεί να αλλάξει κάπως απόχρωση. Εν πάση περιπτώσει είναι η Κομισιόν η οποία έχει ακόμα τη δυνατότητα να αποφασίσει και επίσης ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα του λιμενικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό λαμβάνεται υπόψη στην συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων σε ό,τι αφορά επίση τι βραχίε θαλάσσιε συγκοινωνίε και του αυτοκινητοδρόμου τη θάλασσα, εξακολουθούμε την επεξεργασία μα στην Κομισιόν. Όλα αυτά θέλω να αναφέρω ότι θα περιληφθούν και στον οδικό χάρτη τον οποίο θα παρουσιάσει η Κομισιόν. Ελπίζουμε ότι το έγγραφο αυτό θα δημοσιευτεί μετά από το καλοκαίρι. Οπότε μπορείτε να θεωρείτε ότι το προσχέδιο του είναι ήδη σχεδόν έτοιμο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στις διαβουλεύσεις όπως ήθιστε με όλους τους εμπλεκομένους τομείς, τόσο με την, τις εθνικές αρχές όσο και με τους εμπλεκόμενους της επιχειρήσης και τους ε, εργαζομένους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το οδικός χάρτης Κομισιόν. Απλώς οι κατευθυντήρες γραμμές για την φορολογία δεν θα εμφανιστούν πριν από το 2011 παρά την θέλησή μας. Θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό νωρίτερα, αλλά οι διαδικασίες δεν μας, εμποδίζουν, δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε πιο γρήγορα. Είναι σε δύο στάδια αυτή η διαδικασία. Καταρχήν υπάρχει ένα έγγραφο, ακολουθεί η διαβούλευση με τους εμπλεκομένους και μετά καταλήγουμε στο τελικό έγγραφο της Κομισιόν. Επομένως δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το εκπληρώσουμε. Εν κατακλείδη θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο εισηγητή για την εκθεσή του η οποία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την Κομισιόν και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο και προς τους οποίους μπορώ να πω ότι τα σχόλιά τους θα ληφθούν υπόψη από την Κομισιόν με μεγάλη προσοχή και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Βαντάλε να απαντήσει. Ε, με ρωτάτε ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Τα έχω σημειώσει, αλλά θα ξεκινήσω με μερικές γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, επίτηδες έχω επικεντρωθεί σε κάποια θέματα που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά από πλευράς του Κοινοβουλίου μας. Είναι εύκολο να μιλάμε γενικά για την θαλάσσια πολιτική. Ένα σωρό πράγματα μπορούμε να πούμε, είναι αλήθεια. Αλλά εγώ επίτηδε, περιορέστηκα σε 6-7 θέματα μόνο, γιατί για μένα αυτές οι θεματικέ ενότητε είναι οι σημαντικέ. Όπω είπε ο κ. Φλάκιαστα, ναι, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί για την συνέχεια όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και τη θαλάσσια πολιτική. Επίτηδες επικεντρώθηκα λοιπόν σε αυτά τα θέματα και περιορίστηκα σε 6 με 7 θεματικές ενότητες. Θα μπορούσα να διευρύνω το θέμα, ναι, αλλά σας λέω ότι ήταν συνειδητή επιλογή να περιοριστώ. Τώρα, για να απαντήσω στις συγκεκριμένες σας ερωτήσεις με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο Κουμουτσάκος, που δεν είναι εδώ τώρα, με ρώτησε για την παράγραφο 16. Να εξηγήσω περισσότερο τι εννοώ με την εισαγωγή ενός φόρου επί των καυσίμων στη δεξαμενή. Μα είναι απλό, Πρόεδρε. Ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παράγραφο αυτή να σκεφτεί και να αναζητήσει άλλα εναλλακτικά μέσα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος από την θαλάσσια ναυσιπλοεία και σαν παράδειγμα δίνω την εισαγωγή ενός φόρου επί των καυσίμων στη δεξαμενή. Διότι έχουμε οξύδια του αζότου και οξύδια του θείου και θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφοροποίηση στη φορολόγηση ανάλογα με το αν πρόκειται για καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον ή όχι. διάφοροι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον θα μπορούσαν να μην πληρώνουν φόρο. Ενώ εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν καύσιμα τα οποία είναι επιζήμια για το περιβάλλον να το νιώσουν και στην τσέπη τους. Όλα αυτά βέβαια εμπίπτουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι που είναι η έννοια των πράσινων λιμένων σκάφη τα οποία επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον να πληρώνουν λιγότερο για να πάνε στα λιμάνια αυτά. Ένα σύστημα bonus μάλους δηλαδή. Έτσι δίνουμε κίνητρα στους επιχειρηματίες, εφοπλιστές υπέρ του περιβάλλοντος. Θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο, είπαμε με τη σειρά θέλω να απαντήσω στους συναδέρφους υπάρχει περιθώριο για τροπολογίε. Έτσι, πάντως αυτό που θέλω να πω πάνω απ' όλα είναι ότι υπάρχει το θέμα των ελάχιστων προδιαγραφών όσον αφορά το πλήρωμα. Η εμπειρία μου που είναι μακρά εμπειρία είναι ότι είναι καλύτερα να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει ένα πλήρωμα. Να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Έτσι κι περιμένω ό,τι προτάσεις έχετε να κάνετε, να υποβάλλετε τροπολογίες. Για τον συνάδελφο Τούτσα που είπε ότι με τις σημαίες, ναι, πράγματι, υπάρχει αυτό στην αυσοπλοία, εδώ και πολύ καιρό η αλλαγή σημαίας. Το έχουμε δει αυτό και στην εσωτερική ναυσιπλοεία είχα πει ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε στήριξη σε μέτρα που θα αποφεύγουν το φαινόμενο αυτό και με αυτό συμφωνώ. Τέλος, της συνάδελφο Τικάου. Πράγματι, υπάρχουν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίζα λίστα που τα κατονομάζουμε Αυτό όμως δεν είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν ε, να μην είναι κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κατάλογο αυτό. Στην παράγραφο 22 και 23 της πρότασής μου αναφέρω κάτι σχετικά. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλα σχόλια έχετε να κάνετε, ευχαρίστως να υποβάλλετε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαντάλ. Πρότασή μου είναι 2 Μαρτίου προθεσμία για τις τροπολογίες, 22 Μαρτίου συζήτηση στην ε, Επιτροπή μας ε, και τον και λοιπόν Ολομέλεια τον Απρίλιο. 23 Μαρτίου η ψηφοφορία και Ολομέλεια τον Απρίλιο. Είστε όλοι ευτυχείς, ο εισηγητής συμφωνεί. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για την έκθεσή σας. Επόμενο θέμα στο, στην ημερήσια διάταξη είναι το σχέδιο πρότασης ε, για τους προσανατολισμούς ε, για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων, κυρίως δε για διατύπωση. <laughs> το πήρε ο πρόεδρος, δηλαδή εγώ, γιατί κανείς άλλος δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται και να το θέλει, εν πάση περιπτώσει. Εδώ έχουμε μια σειρά τροπολογιών, όμως θα ήθελα πρώτα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή μας ε, ότι συμφωνήσαμε την τελευταία φορά ότι θα, θα προσπαθούσαμε να έχουμε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης επ' αυτού. Δεν πρόκειται για αναδιατύπωση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, απλώς αφορά διόρθωση κάποιων τεχνικών λεπτομεριών ε, που διορθώνονται σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Ε, υπάρχουν λοιπόν και κάποιες τροπολογίες ε, οι οποίες ε, απλώς θέλησαν να επιφέρουν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά, τροποποίηση όσον αφορά τους χάρτες και τα ονόματα και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι κατά της οποιασδήποτε τροποποίησης των διευρωπαϊκών δικτύων. Όμως να σας πω το εξής, για να μπορέσουμε να περάσουμε ε, την πρώτη ανάγνωση, να ψηφίσουμε από των δύο τροπολογιών με τις οποίες ε, συμφώνησαμε το Συμβούλιο και δεν έχουμε πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Οι ε, τροπολογίες μου αφορούν αφενός την ενδυνάμωση της θέσης της Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή, την Επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή και την ανάπτυξη των προσανατολισμών κτλ. Και τη δεύτερη τροπολογία ε, αφορά τον, ε, τη χρονολογία, τον στόχο ε, και τον αριθμό των χωρών. Η αρχική μου δεύτερη τροπολογία απεσήρθη διότι φαίνεται ότι υπήρξε ένα νομικό πρόβλημα με την διατύπωση και ε, εν πάση περιπτώσει τώρα η νέα διατύπωση έγινε δεκτή από το Συμβούλιο το οποίο είχε ενστάσει όσον αφορά την πρώτη διατύπωση. Έχουμε λοιπόν ε, τις δύο μου τροπολογίες ε, και με τις τροπολογίες αυτές γίνεται δεκτή και η πρόταση τροποποίησης του Συμβουλίου. Έχουμε επίσης τροπολογίες από την κυρία Κρέμες και τον κύριο, ο κύριο και την κυρία Λίχτεμπεργκ. Ε, πρόκειται πάντα για τροπολογίες οι οποίες αφορούν την προσθήκη των χαρτών και εν πάση περιπτώσει αν θέλετε εσείς να τροποποιήσετε τους χάρτες μπορείτε να το κάνετε αλλά ο σωστός τρόπος και χώρος για να αναθεωρηθούν και να διορθωθούν οι χάρτες είναι όταν θα προταθεί η αναδιατύπωση της πραγματικής οδηγίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Γι' αυτό λοιπόν θα, περί, θα πρότεινα να ε, περιμένουμε μέχρι τότε έτσι ώστε να προτείνεται οποιαδήποτε τροποποίηση. Υπάρχει και άλλη μια πρόταση της κυρίας Τικάου, αιτιολογική σκέψη 20, με την οποία δεν συμφώνησε το Συμβούλιο και που ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσε να δυναμητήσει τη συμφωνία επί πρώτης ανάγνωσης. Γνωρίζω ότι η κυρία Τικάου θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Όμως εγώ πιστεύω ότι με την αλλαγή του κειμένου του 2007 καλύφθηκαν ε, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Όταν έγιναν λοιπόν οι απαραίτητε τροποποίησει και προσαρμογές του κειμένου μετά από την ένταξη των ε, χωρών ε, αυτών ε, διορθώθηκε το κείμενο και δεν υπάρχει πλέον κείμενο και πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει και εγώ στην τροπολογία μου 2 έχω αναφέρει ότι θα πρέπει να βρίσκονται οι χάρτες των 10 κρατών μελών που αναφέρονται στην πράξη προσχώρησης του 2003. Προτείνω λοιπόν να παραμείνουμε στις δύο τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής έτσι ώστε να περάσουμε στην πρώτη ανάγνωση. Ε, ε, ε, καταλαβαίνετε ότι εάν αποτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια τότε θα πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση και πιστεύω ότι έτσι θα δυναμητήσουμε αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό, δηλαδή η αναδιατύπωση της, των ίδιων, της ίδιας οδηγίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεμπερδεύουμε με αυτό τώρα. Έχω τον κύριο ε, Πακέ και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω να προσθέσω το οτιδήποτε εκτός από την ευγνωμοσύνη που νιώθω για το έργο σας ως εισηγητού και το έργο της Επιτροπής σας και για την προσπάθεια σας να επιτύχουμε σε μια συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Αυτή η αναθεωρημένη πρόταση δημιουργεί πράγματι μια ενιαία βάση για τη μεταρρύθμιση και από την άποψη αυτή θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η εκθεσή σας για να υπάρξει η μεταρρύθμιση της πολιτικής μας και η επιτυχία μιας συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης θα ήταν πάρα πολύ θετική για τη διαδικασία και για την ουσία των τροπολογιών Ξέρω ότι υπάρχει για πολλές από αυτές τις τροπολογίες συμφωνία του Συμβουλίου. Υπάρχει όμως κάποιος κίνδυνος για ορισμένες τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν τύχει συμφωνίες από το Συμβούλιο και νομίζω ότι εάν εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σωστή αντιμετώπιση για τις υπόλοιπες τροπολογίες της Επιτροπής σας, αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Είπα 8 συν 2, εννοούσα μάλλον 10 συν 2 για τα νέα κράτη-μέλη. Κύριε Κάντσιεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό. Και πραγματικά περιμένω να κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας για το θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι για την Επιτροπή μας εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως είπατε όμως και εσείς, το κείμενο που μας απασχολεί σήμερα είναι καθαρά τεχνικής φύσης και επομένως ε, η ευρυνή ψηφοφορία θα αποτελέσει ε, την εκκίνηση της ε, συνολικής επαναδιαπραγμάτευσης των ΤΕΝΣΑ για τα επόμενα χρόνια. Λίγες λοιπόν είναι οι τροποποιήσεις βάσει των τροπολογιών που έχετε υποβάλει. Τις θεωρώ σκόπιμες και χρήσιμες έτσι ώστε να επιτύχουμε ένα σωστό και συνεκτικό τελικό κείμενο. Ε, στηρίζω λοιπόν τις ε, τροπολογίες σας και δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος γιατί δεν είναι ακόμα ο χρόνος να ασχοληθούμε με τα θέματα τα οποία προτείνουν οι άλλοι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους. Νομίζω ότι το κύριο μέλημά μας θα είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Το κείμενο έχει κωδικοποιηθεί, πρέπει να κωδικοποιηθεί σε πρώτη ανάγνωση έτσι ώστε να επιτραπεί ή ε, ο επαναπρογραμματισμός των διευρωπαϊκών δικτύων που είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Και ελπίζω ότι όταν θα ε, μπούμε στη συζήτηση επί της ουσίας. Ε, μέσω σωστής συζήτησης θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια χωροθέτηση σωστή, προγραμματισμένη, ε, διατροπική γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης εξίσου σημαντικό θεωρώ ο, ο προγραμματισμός αυτός να ακολουθείτε ε, από τις προσπάθειες της Επιτροπής ε, και του, ε, Συμβουλίου για τη δημιουργία ταμείου για την χρηματοδότηση μεμονωμένων προγραμμάτων. Ευχαριστώ κύριο Στέρξ. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζω την πρόταση που κάνατε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα που υπάρχει ενώπιόν μας. Εγώ υποστηρίζω τις τροπολογίες της σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπορούμε να φανταστούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν η φαντασία μας έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Πριν από 5 ή 7 χρόνια είχαμε 10 κράτη-μέλη λιγότερα. Αλλά αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο σε σχέση με αυτό το έγγραφο. Εμεί θα πρέπει να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 27 κράτη-μέλη της σήμερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μικρές τροποποιήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νέα κράτη-μέλη και έχουμε φτάσει πια στα 27 κράτη-μέλη. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αφορά την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, υποστηρί... να λαμβάνει υπόψη και τα 27 κράτη-μέλη. Γι' αυτό υποστηρίζω τι προτάσει τη κυρία ε, Τίκαου. Η τεχνική τώρα μαγνητική αιώρηση. Έχω συζητήσει με τον Βίλι Πίτσικ, ο οποίο δυστυχώ δεν είναι πια μαζί μα και ήταν σαφέ ότι ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπήρξε κάποια υποστήριξη της του Transrapid, δηλαδή των τρένων που χρησιμοποιούν τη μαγνητική αιώρηση. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη μέσα από διάφορες τεχνικές σηματοδότησης, μέσα από τέσσερα διαφορετικά πλάτη γραμμών, να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο σύστημα σιδηροδρομικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν απαραίτητο λοιπόν και είναι σύμμορφο με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε τονίσει κατ' επανάληψη ο Βίλι Πίτσικ. Διότι εάν οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν ένα σύστημα το οποίο δεν είναι συμβατό με τα άλλα, αυτό δεν έχει να κάνει με μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Ακόμα και η τωρινή γερμανική κυβέρνηση δεν λέει πια τίποτα για το Transrabbit μέσα στο πρόγραμμά της. Ούτε στην Βαβαρία όπου είχε προταθεί αυτό. Δεν ξέρω λοιπόν αν εμείς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό. Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να βρούμε σε οποιαδήποτε κοινή θέση. Ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της γραφειοκρατίας λέγεται Στόιμπερ και ήταν ο Πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βαβαρίας στο παρελθόν και ο οποίος τότε είχε υποστηρίξει τον Transrapid. Και ήταν σαφές εκείνη την εποχή ήδη ότι 80% του πληθυσμού δεν υποστήριζε το Transrapid, το σχέδιο αυτό εκείνη την εποχή. Γιατί λοιπόν ξαναγυρίζει αυτό το πράγμα που κανεί δεν το θέλει, αυτό για μένα είναι ένα έρηγμα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί εμεί δεν βρισκόμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να επανέλθω σε αυτά τα οποία λέει η κυρία Τικάου. Πρέπει να σκεφτούμε σαν μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών και όχι σαν παράγματα διαφορετικών κρατών που έχουν διαφορετικές πολιτικές στον τομέα των μεταφορών. Κυρία Τικάου και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι όλοι κατανοούμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε μία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Πρέπει όμως να σας πενθυμίσω ότι η τροπολογία μου υπαριθμών 6 και η τροπολογία μου υπαριθμών 5 ασχολούνται με τεχνικά ζητήματα αυτό δεν αλλάζει το περιεχόμενό τους. Να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι και οι δύο τροπολογίες έχουν μεν τεχνικό χαρακτήρα, αλλά θέλουν να διορθώσουν τα ασφάλματα τα οποία υπήρχαν σε προηγούμενα έγγραφα. Έρχομαι στην τροπολογία 5 καταρχήν. Συγγνώμη, στην 4, στην ε, δική σας τροπολογία κύριε Πρόεδρε, λέτε εσείς κάτι το οποίο επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με την τροπολογία 5. Είναι σχεδόν ταυτόσιμες, αλλά η διαφορά είναι ότι αναφέρεται μονάχα η προσχώρηση, η συμφωνία προσχώρησης για κράτη που μπήκανε μετά το 2003. Θα μπορούσε ίσως κανείς να τροποποιήσει την τροπολογία 4 που να λαμβάνει υπόψη και τα τελευταία κράτη, για τη Ρουμανία δηλαδή και τη Βουλγαρία που ε, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 και η αντίστοιχη συμφωνία ελήφθη το 2005. Το έτος 2010, δηλαδή σήμερα εμείς θα πρέπει να εγκρίνουμε ένα έγγραφο το οποίο θα είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρακάμψουμε το γεγονός ότι έχουν εισέλθει δύο διαδοχικά κύματα κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στον κανονισμό 2006 υπάρχει η έμεση αναγνώριση της διεύνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εφόσον τώρα επικαιροποιούμε αυτό το νομοθέτημα, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη πλήρως την ε, ε, διεύνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωρίσουμε τις απόρριες αυτής της ε, διεύνησης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ πιστεύω ότι το Συμβούλιο στα πλαίσια της κοινή λογικής θα δεχτεί αυτές τις τροπολογίες. Για τροπολογία υπαριθμών 6 εδώ έχει τροποποιηθεί ο τίτλος. Αφορά τα θέματα της Μαύρης Θάλασσας. Καταρχήν αφορούσε τα θέματα όλης της Μαύρης Θάλασσας, τώρα περιορίζεται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά για τη Μεσόγειο, για τη Βαλτική, είναι σημαντικό να έχουν οι χάρτες τη σωστή ονομασία. Επομένως και στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας θα πρέπει να δοθεί ένας σωστός τίτλος, το οποίο δεν είναι μόνο Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά Μαύρη Θάλασσα, εύξηνος πόντος. Γι' αυτό έχω καταθέσει αυτές τις δύο τροπολογίες που εγώ πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στην κοινή λογική και ελπίζω ότι θα την υποστηρίξετε αγαπητοί συνάδελφοι. Απαντώντας σε αυτά που είπατε, ήθελα να πω ότι για την τροπολογία 4, αν διαβάσετε αυτά τα οποία λέω, υπάρχει μια πολύ σημαντική φράση που λέει όλα τα κράτη-μέλη. Επομένως όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπεριληφθούν εάν εγκριθεί αυτή η τροπολογία. Η ιδέα αυτή ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν συμπεριλαμβάνονται αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το απορρίπτω γιατί εγώ αναφέρομαι σε όλα τα κράτη-μέλη οπότε αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόζει τον κανονισμό σε όλα αυτά τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα κράτη σε, στη μνήα όλα τα κράτη. Δεν μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι όταν λέμε όλα δεν καλύπτει τα 27 κράτη-μέλη. Επομένως εγώ με κάθε σεβασμό παραμένω στην δική μου διατύπωση. Κύριος Κράμερ χωρίς ε, μικρόφωνο. 15 και 10 κάνει 25 και όχι 27 λέει ο κύριος Κράμερ. Μα Μάικελ, όταν λέμε όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή είναι 27 κράτη-μέλη. Μα στη μετάφραση λέει 15 συν 10. Λοιπόν, να μην κάνουμε διάλογο τώρα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο κάναμε αυτή την τροποποίηση και υπήρξε μεγάλη προσοχή και σε νομικό επίπεδο και σε πραγματολογικό επίπεδο ώστε να καλύπτονται όλα τα κράτη-μέλη. Και πιστεύω λοιπόν με την τροπολογία μου καλύπτεται και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Μα και η Βουλγαρία και η Ρουμανία στο Συμβούλιο των Υπουργών έχουν συμφωνήσει με μια τέτοια διατύπωση. Πού είναι το πρόβλημα για την τροπολογία τώρα που αφορά τη Μαύρη Θάλασσα. Είμαι εναντίον, γιατί αλλάζει μια γεωγραφική έννοια. Αντί να μιλάμε για Βουλγαρία και Ρουμανία, μιλάμε για τη Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα καλύπτει και άλλες χώρες πέραν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα στην επόμενη μεταρρύθμιση των διευρωπαϊκών δικτύων να αλλάξουμε την ονοματολογία. Δεν έχω πρόβλημα να βγάλουμε την ε, μνήα του Transrapid από, τη, τα από την ε, μεταρρυθμισμένη μνήα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και συμφωνούσα απόλυτα με τον Βίλιτσι Πίτσεκ αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει σε αυτή την έκθεση. Πρέπει να γίνει στην έκθεση για τη μεταρρύθμιση των διευρωπαϊκών δικτύων. Εγώ υποστηρίζω όσο μπορώ περισσότερο τη θέση που έχετε, αλλά δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή την ε, τροποποίηση. Είπατε ότι το τράζαπι δεν έχει καμιά σχέση με την Ευρώπη και τις μεταφορές. Ναι, αλλά δεν έχει και καμιά σχέση αυτή η τροποποίηση που θέλετε να κάνετε με αυτή την έκθεση. Τώρα, για να προσθέσουμε στην τροπολογία 4 και το 2005, το δέχομαι. Αν όμως υπάρχει σαφήνεια με μια προφορική τροπολογία ότι αυτό είναι σωστό σε νομικό επίπεδο και είχαμε πολλά προβλήματα σε νομικό επίπεδο και αν το Συμβούλιο το δεχτεί αυτό το πράγμα, εγώ μπορώ να προσθέσω 2003 και 2005 στο κείμενο για τις ημερομηνίες που αποφασίστηκε η προσχώρηση περαιτέρω κρατών. Αλλά θέλω σαφήνεια για αυτό το θέμα πρωτού ψηφίσουμε. Και αν λοιπόν δεν έχουμε πρόβλημα, θα δεχτώ αυτή την προφορική ερώτηση. Αν μου πούν όμω τώρα ότι σε νομικό επίπεδο είναι προβληματική, εγώ θα πρέπει να παραμείνω στην αρχική μου τροπολογία. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύα, γρήγορα. Μια μικρή ερώτηση. Δεν αφορά. Αφορά μάλλον το θέμα Βουλγαρία, Ρουμανία και Μαύρη Θάλασσα επειδή δεν μιλάμε για κράτη-μέλη αλλά για γεωγραφικές περιοχές. Είναι πιο σωστό να μιλάμε για μαύρη θάλασσα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία είναι αρμόδια για αυτή την περιοχή. Είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία και όχι η ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει η των δύο αυτών κρατών μελών που έχουν παρουσία στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Για το 2005 δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό. Αλλά για την περίπτωση αυτή δεν ξέρω αν θα αυτό θα γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να το ελέγξω σε νομικό επίπεδο. Ε, και μπορούμε τότε σε αυτή την, ε, την περίπτωση να το αλλάξουμε. Αλλά όσον αφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σαν αναφορές ε, για τον εύξηνο πόντο, εγώ δεν συμφωνώ. Και εν πάση περιπτώσει έτσι ήταν και στο αρχικό κείμενο των ΤΕΝΣ. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή αν ήταν λάθος και δεν είναι, δεν είναι δουλειά αυτή τη έκθεση να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Αυτό που μας απασχολεί εδώ σήμερα είναι μια τεχνική έκθεση η οποία αφορά κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν στα αρχικά τένς έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ησυχία μας σε περαιτέρω μεταρρύθμιση ε, των τένς που πραγματικά είναι πολύ απαραίτητη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα γρήγορα να ελέγξουμε εάν είναι δυνατόν να αλλάξουμε το 2003 να τον αντικαταστήσουμε με το 2005, εάν αυτό από νομικής απόψεως δηλαδή είναι ε, σωστό και στέκει. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα μας πούν για μία ακόμα φορά δεν υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου για το 2005. Mm, Σίλβια, πρόεδρος. Ξέρεις ότι με μεγάλη συμπάθεια ακούω αυτά που λες, αλλά δεν πρέπει να ξεχανάμε ότι εδώ έχουμε τεχνικές λεπτομέρειες και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβια όσον αφορά τον τίτλο του εύξηνου πόντου. Εάν δείτε αν δει κανείς τον ε, χάρτη της Μεσογείου, διαπιστώνει ότι παρότι υπάρχουν εκεί χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ο χάρτης με επικεφαλίδα ε, ε Μεσόγειος Επομένως υπάρχει πρόβλημα με τον χάρτη παριθμών 5,6. Είτε τώρα είτε μετά θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον, την επικεφαλίδα του χάρτη αυτού. Γιατί να μην το κάνουμε λοιπόν τώρα. Όσον αφορά τώρα την πράξη προσχώρησης του 2005. Υπάρχει μια αρχή ε, με την οποία εγώ συμφωνώ, δηλαδή ότι θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι πράξεις προσχώρησης. Και όταν θα έχουν τροποποιηθεί οι χάρτες, τότε οι αλλαγές θα γίνουν σύμφωνα ε, με τις ε, τελευταίες χώρες οι οποίες θα έχουν προσχωρήσει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα ε, στην αναφορά της πράξης του 2005, γιατί απλώς αναφέρουμε και τις δύο τελευταίες πράξεις προσχώρησης. Πρόεδρος, απήντησα ήδη το θέμα του 2003 και 2005. Τώρα, όσον αφορά την Μεσόγειο, δεν μπορώ να το αλλάξω γιατί έτσι είναι η επικεφαλίδα σε αυτό το χάρτη στην παρούσα έκθεση. Ε, ενώ για τον χάρτη του εύξηνου πόντου το 5,6 αναφέρεται ως Βουλγαρία-Ρουμανία. Δεν μπορώ λοιπόν να αλλάξω. Αυτά έχω, με αυτά θα μείνω. Δεν μπορώ να αλλάξω αυτά τα ονόματα για την ώρα. Πρόκειται για μία ακόμα φορά σας το λέω, για μία τεχνική έκθεση η οποία η οποία έχει στόχο την τεχνική διόρθωση κάποιων λεπτομεριών δεν ξέρω, πέστε μου κι εσείς κάτι. Προσπαθώ εδώ να πω απεγνωσμένα και το επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για αναδιατύπωση της οδηγίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πρόκειται για μία, ε, ε, ε, για, πρόκειται για κάποιες τροποποιήσεις τεχνικές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Ε, Κομισιόν, δεν μπορώ να ε, πω τίποτα πιο πιστικό από όλα αυτά που είπατε εσείς. Ε, τώρα όσον αφορά την τροπολογία 4, να πούμε το εξή. Η, η αιτιολογική σκέψη 20 δεν λέει ότι έχουμε 5, 10, 15 ή 20 χάρτες. Αναφέρει ότι έχουμε τώρα ένα νέο παράρτημα με όλες τις χώρες μέλη. Και μετά υπάρχει και η φράση η οποία αναφέρεται στην πράξη ε, προσχώρησης ε, του 2000 και αναφέρεται ότι το όλο εγχείρημα έχει στόχο να τροποποιηθούν, να διορθωθούν μάλλον κάποια λάθη τα οποία είχαν ε, παρισφρήσει στο κείμενο με την πράξη ε, προσχώρησης του 2003. Επομένως εδώ δεν γίνεται λόγος παρά μόνο για τις τεχνικές διαδικασίες, ούτε για, την ίδια την έννοια των διευρωπαϊκών δικτύων, ούτε για οποιαδήποτε αναδιατύπωσή τους ή μεταρρύθμιση τους. Νομίζω ότι είναι ένα καθαρά πρακτικό θέμα. Όσον αφορά τις δύο άλλες τροπολογίες, ε, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας ότι όλα αυτά τα ουσιώδη ζητήματα θα πρέπει να συζητηθούν στην πραγματική συζήτηση που θα γίνει για την ε, ε, στρατηγική των ευρωπαϊκών δικτύων. Εκεί θα μιλήσουμε για μεθοδολογία, εκεί θα έχουμε βεβαίως ε, και την διαβούλευση της Επιτροπής που θα ξεκινήσει τον την Άνοιξη και τότε θα έχουν όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας χώρο και χρόνο για να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, εσεί θα πάρετε τις αποφάσεις σας, ε, μπορείτε να τη δεχτείτε την πρότασή μου, την ξέρετε την πρότασή μου, ξέρετε την άποψή μου. Αύριο θα έχετε την ε, ψήφο σας με την οποία θα συμφωνήσετε ή θα διαφωνήσετε. Ε, θα σου δώσω ακόμα μια λόγο γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, αλλά να είσαι σύντομη. Από ό,τι κατάλαβα, η Επιτροπή η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στην πράξη προσχώρησης του 2005. Όμως αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ε, αντίθετη νομική άποψη για τη συμπερίληψη της ε, πράξης προσχώρησης του 2005. Επομένως θα πρέπει να γίνει κάποια αναφορά στην τελευταία πράξη προσχώρησης. Πρόεδρος, ε, εντάξει, ε, μπορούμε να πούμε ότι θα, ε, και με την πράξη προσχώρηση του 2005 διορθώνουμε τα λάθη της πράξης προσχώρησης του 2003. Πάρα πολύ ωραία. Um, Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, έκθεση Κούν σχετικά με την περιφέρεια της Βαλτικής θάλασσας. Θα ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο να πάρει τη θέση μου εδώ για λίγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε γνωμοδοτούσα επιτροπή ως Επιτροπή Μεταφορών για την πολιτική που αφορά την Βαλτική και εγώ ως εισηγητής θα ήθελα να περιοριστώ σε θέματα μεταφορών. Είναι δέκα σημεία τα οποία έχω επεξεργαστεί. Προφανώς είναι η βασική αρτηρία της περιοχής της Βαλτικής η διαδρομές θαλάσσιων μεταφορών και πρέπει να παραμείνουν βασική αρτηρία και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις συνθήκες εκεί. Επίσης τα οι ευρωπαϊκά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο και χώρες όπως η Νορβηγία και η Ρωσία παίζουν σε αυτά και σημαντικό ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να συμπεριλάβουμε πλήρως τη Βαλτική στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η ήδη υφιστάμενη υποδομή, είτε είναι σιδηροδρομική, είτε είναι οδική, είτε αφορά εσωτερικούς υδάτινου δρόμους, θα πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αυτό ήταν κάτι που συζήτησαμε όλου όλους τους συζητητέ και αυτό ήταν κάτι που όλοι θεωρήσαμε ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμφωνήσαμε επίση ότι είναι απαραίτητο η μεγάλη άξονες μεταφορές όπως ο διάδρομος 1 από το Παλέρμο στο Βερολίνο να επεκταθεί και στην περιοχή της Βαλτικής. Και επίσης ο θαλάσσιος δρόμος 21 και η Ρέα Μπάλτικα που είναι το, το ένα και η Ρέα Μπάλτικα είναι, η είναι ε, συνδρομική άξονες. Θα πρέπει να ληφθούν και αυτοί οι υπόψη. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι ήδη υπάρχοντες διάδρομοι φτάνουν στη Βαλτική και επίσης να λάβουμε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος η οποία μπορεί να θυγεί από την επέκταση αυτών των διαδρόμων. Θέλουμε να υπάρξει λοιπόν η ανάπτυξη των μεταφορών και των διαδρόμων μέχρι τη Βαλτική, αλλά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Επίση, η στρατηγική της Βαλτικής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική ε, δυνατότητα βραχαίων θαλασσίων μεταφορών αυτό είναι μια σωστή στοχοθεσία, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια για τα καύσιμα τα οποία θα χρησιμοποιούνται να μην είναι τόσο αυστηρά ώστε να έχουμε στρεβλωτικό αποτέλεσμα ώστε να μετακυλιστεί, να μεταφερθεί η εμπορευματική κίνηση από τις θαλάσσιες μεταφορές λόγω των υψηλών προδιαγραφών στα καύσιμα πάλι στους, στους οδικές μεταφορές. Η ασφάλεια επίσης παίζει μεγάλο ρόλο στη θάλασσα και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις πτυχές οι οποίες επηρεάζουν και τον τουρισμό. Περιοχές, παραδείγματο χάρη, στενών θαλασσίων περιοχών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό, το πρίσμα της δημιουργίας σταθμών ραντάρ που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών εκεί ενώ συγχρόνως όμως θα πρέπει να έχουμε και την πρέπουσα προσοχή στις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν για το περιβάλλον και για τον τουρισμό. Επίσης, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας, τα θέματα λοιπόν αυτά τουρισμού, το φόρουμ του τουρισμού στην Βαλτική έχει υπογραμμίσει την ιδιαίτερη δυνατότητα Τη ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή αυτό, αλλά προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι μια καλύτερη προσβασιμότητα της ε, Βαλτική, ώστε να μπορούν αυτοί οι οποίοι κάνουν μονάχα σύντομε διακοπέ να έχουν τη δυνατότητα ταχαίω να φτάσουν σε περιοχέ τη Βαλτική που θεωρούν ελκυστικέ για τουριστικέ δραστηριότητε. Όλοι αυτοί είναι λοιπόν στόχοι του οποίου εμεί θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε για την πολιτική μεταφορών στη Βαλτική, ώστε να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Βαλτικής χάρη σε καλύτερη παροχή μεταφορικών συνδέσεων με την περιοχή της Βαλτικής ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αηφόρο ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. Αυτός ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κούν, Αγαπητοί συνάδελφοι, και ο σκιώδης εισηγητής μας είναι κάπου στο δρόμο από την Λιθουανία στις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ λοιπόν να τον αντικαταστήσω πλήρως, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα μπορώ να δώσω δίκαιο σε ορισμένα σημεία τα οποία υπεγράμισε. Αναφερθήκατε κι εσείς στο, στα σημεία αυτά 5 και 6 ε, και σίγουρα εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προβληματική για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από τα καύσιμα των ε, πλοίων και θα πρέπει να προσέξουμε ότι οι προδιαγραφές όπως είπατε για την ε, περιεκτικότητα σε θείο δεν θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρές που να μεταφερθεί η κίνηση των ε, εμπορευμάτων στην, ε, στις μεταφορέ μεταφορές και όχι στη θάλασσα. Ο κύριος Βανδάλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς ε, αυτός από εμά που ασχολείται περισσότερο με αυτά τα θέματα δεν είναι παρόν. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κάποια σχόλια, αλλά κατά τα άλλα θα υποβάλουμε τροπολογίες. Μιλήσατε για 10 σημεία, όντως είναι τα πιο σημαντικά, πράγματι. Όμως, πρέπει να αναρωτηθούμε όσον αφορά την σχέση των βαλτικών χωρών με την Ρωσία. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκονται δίπλα, υπάρχουν θέματα τελωνιακών διατυπώσεων, υπάρχουν επίσης πτυχές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη των βαλτικών χωρών. Η απομόνωση, επίσης, το είπατε σωστά, το υπογραμμίσατε, ότι οι βαλτικές χώρες, ότι για αυτές τις χώρες τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γενικά πάντως, εντάξει, καλή προσέγγισή σας, συμφωνούμε, αλλά θέλουμε πιο πολλέ διευκρινήσει. Οπότε οι τροπολογίε μα θα πηγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση, θα είναι πιο συγκεκριμένε. Ευχαριστούμε, κύριο Κράμερ, έχει τον λόγο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κούν για την έκθεση αυτή και για το γεγονό ότι έχει συγκεντρώσει την προσοχή του στα σημαντικότερα θέματα. Φυσικά, συμφωνούμε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ Βερολίνου με την Βαλτική. Αλλά αν βλέπετε σε εφημερίδες ότι αναφέρεται ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στηριοδρομικές υποδομές στον τομέα αυτό μεταξύ Βερολίνου και Βαλτικής, αυτό είναι και το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ελκυστική τη δημιουργία σιδηροδρομικών ε, μεταφορών. Επίσης, η σύνδεση με την Σκανδιναβία μέσω της ε, Δανίας και μέσω του Αμβούργου και η σύνδεση μέσω Ρόστοκ δεν πρέπει να τύχει να την ε, παραμελήσουμε. Παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση σωστή με τις γέφυρες οι οποίες οδηγούν στην Δανία από τη Γερμανία. Επομένως πολλές φορές κάνουμε αυτές τις ενέργειες, δημιουργούμε υποδομές με γέφυρες χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη και το γεγονός να υπάρξει σύνδεση με συνδρομικές μεταφορές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν αυτή την λογική. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τους άξονες μεταφορών, γιατί γνωρίζουμε ότι τα κράτη της Βαλτικής έχουν πολλά προβλήματα οι Λιθουανοί λένε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν το θέλουν οι Πολωνοί. Οι Λετονοί λένε θέλουμε να φτιάξουμε αλλά δεν το θέλουν οι Λιθουανοί και μετά οι Πολωνοί έχουν πρόβλημα με τους Λετωνούς. Όλα αυτά είναι πραγματικά ενοχλητικά. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλιστεί ότι θα ξεπεραστούν αυτές οι διαφορές και θα υπάρξει η απαραίτητη σύνδεση των κρατών αυτών με την ενδοχώρα τους. Αλλά ξέρουμε ότι ο άξονας Υ, Ανόβερο, Αμβούργο, και Βερολίνο, εκεί είναι ένας άξονας όπου μπορούμε να επιταχύνουμε τις ε, μεταφορές, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τα σημεία τα κομβικά. Δηλαδή σημεία όπως ε, η Βρέμη, το Αμβούργο και το Ανόβερο θα πρέπει να εξυγχρονιστούν για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις γέφυρες που οδηγούν στη Δανία και τον άξονα Υψηλό. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μία σταθεροποίηση <clears throat> των ε, ήδη υπαρχόντων σιδηροδρομικών αξιών και να υπάρξει και φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση με τους λιμένες μέσω σιδηροδρόμου. Ευχαριστούμε. Κύριε Κράμερ, εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν υπάρχει από ό,τι έχω καταλάβει, ούτε καν άλλο ζητάει το λόγο για την έκθεση αυτή. Πρόβλημα υπάρχει γιατί ακόμα και οι σκιώδε ε, είναι απόντες, οπότε ας απαντήσει λοιπόν ο κύριος Κιούν. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξη που μου έχουν δώσει σε ό,τι αφορά την λεγόμενη αυτή μακροπεριοχή της Βαλτικής. Είναι σαφής λοιπόν η άποψη που έδωσε ο κύριος Φλέκενστάιν για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των θαλασσίων μεταφορών στη Βαλτική έναντι των οδικών μεταφορών. Είναι σαφές κύριε Βαντάλε ότι είναι μια σχετικά κλειστή θάλασσα η Βαλτική σε ό,τι αφορά τις ε, των θαλασσίων μεταφορών. Αλλά από εκεί μπορούν να ξεκινήσουν διαφορές, διαδρομές οι οποίες καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές κρουαζιέρες οι οποίες πηγαίνουν στην περιοχή αυτή. Έχουμε σημαντικές ροές πετρελαιοφόρων που φεύγουν από τη Ρωσία και πηγαίνουν στο Ατλαντικό. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη κύριε Κράμερ και δεν έχουμε καμία απολύτως ε, διαφορά μεταξύ μας απόψεων όταν λέμε ότι είναι απαραίτητο να φτάσουν οι άξονες των διευρωπαϊκών δικτύων μέχρι την Βαλτική. Δεν μπορώ τώρα να περάσω σε λεπτομέρειες στην δική μου ε, γνωμοδότηση γιατί είμαστε μια γνωμοδοτική επιτροπή. Είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή που έχει την ευθύνη να διεξέλθει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εμείς όμως μπορούμε να τονίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση, να είμαστε φιλικοί και προς το περιβάλλον διότι πρόκειται για μια τουριστική περιοχή, μια τουριστική μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν τον λόγο. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα λίγο και ήθελα να πω το εξής. Να προτείνω στον εισηγητή σχετικά με αυτήν την ε, αναφορά για, τον, ε, για την διασύνδεση των αυτοκινητοδρόμων ε, με την Βαλτική. Εγώ πιστεύω ότι ο 23 είναι πάρα πολύ σημαντικό που φτάνει στο Ξδάνσκ να φτάσει τελικά μέχρι και την Βαλτική, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια διασύνδεση μεταξύ Μεσογείου στην ουσία και Βαλτική. Προέδρο, πάρα πολύ ωραία. Να σας δώσω και το χρονοδιάγραμμα σχετικά με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. 2 Μαρτίου οι τροπολογίες, συζήτηση των τροπολογιών στις 22 Μαρτίου στην Επιτροπή, ψηφοφορία πάντα στην Επιτροπή Μεταφορών 23 Μαρτίου και η ψηφοφορία της ίδιας εκθέσεως στην ε, ε, Περιφερειακή Επιτροπή 26-27. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Η κυρία Αγέλα Σέντερ δεν είναι εδώ, η οποία είναι υπεύθυνη για την γνωμοδότηση αυτή. Θα ζητήσουμε ενδεχομένως τον κύριο Κράμερ, ο οποίος έχει ήδη υποβάλει και κάποια τροπολογία. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για την απαλλαγή. Και έλεγα ότι η συγγήτρια δεν είναι εδώ. Αλλά ο κύριος Κράμερ έχει μια τροπολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη η τροπολογία και οι άλλες τροπολογίες άλλωστε. Δεν υπάρχουν άλλες. Ε, μία τροπολογία Κράμερ και η τροπολογία της κυρίας ε, Σέντερ. Αύριο θα ψηφιστεί η γνωμοδότηση. Αυτή δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε επίσης απαλλαγές όσον, απαλλαγές όσον αφορά τους οργανισμούς. Ούτε εδώ υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Έχουμε την επαλλαγή για, το, για την εταιρεία Σεζάρ. Yes. Ε. Θα μιλήσετε γενικά για τις απαλλαγές όλες. πάρα πολύ ωραία. <laughs> Ευχαριστώ. Πολλοί από εμά δυσκολευτήκαμε με τις πτήσεις σήμερα. Γι' αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις. Όντως, πρόκειται για την απαλλαγή. ΕΜΣΑ και ΆΣΑ, Επιτροπή και Εκτελεστικοί Οργανισμοί, το ΣΕΣΕΡ. Και ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες τροπολογίες Όσον αφορά το έμψα είναι η κυρία Σέντερ που έχει υποβάλει ορισμένες τροπολογίες υπογραμμίζοντας τους οργανισμούς με συγκεκριμένα μέτρα και υποστηρίζω τις τροπολογίες της 1 και 2. Όσον αφορά την πολιτική αεροπορία, υπάρχουν άλλες τροπολογίες. Υπάρχουν και μερικές καινούργιες δικές μου. Όπου μιλάω για τις μεγάλες μεταφορές και τις δυσκολίες στο σχεδιασμό όσον αφορά το προσωπικό. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, δυσκολίες γενικής φύσεως. Αναφερόμαστε εδώ στις διοργανικές ομάδες εργασίας που φτιάχτηκαν για τους οργανισμούς προκειμένου η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να μπορούν μαζί και να συζητάνε αυτά τα θέματα. Η κυρία Σέντερ υποβάλλει λίγο πολύ τις ίδιες τροπολογίες με συγκεκριμένο σχεδιασμό, λεπτομερή και συμφωνώ με τις τροπολογίες αυτές. Ο κ. Μπαλσίτης επίσης μιλάει για στόχους και δίκτες σχετικά με τα αποτελέσματα και συμφωνώ και με αυτή την τροπολογία, αριθμός 5. Τώρα για τον οργανισμό σιδηροδρόμων εδώ. Ναι. Υπάρχουν δύο τροπολογίες που εγώ προσωπικά δεν θα τις υποστηρίξω. Γιατί εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω περισσότερο να διευκρινιστεί το θέμα των δύο χώρων που τελικά θα βρίσκεται ο οργανισμός. Αναγνωρίζω ότι στην τροπολογία αριθμός 1 προσπαθείτε να βρείτε κάποια συμβιβασμό. Το αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω ότι προκαλείται επιπλέον κόστος. Ε, τροπολογία είναι τώρα για το ΣΕΣΑΡ του κ. Μπαλσίτη. Άκουσα ότι αποσύρθηκε. Οπότε τελικά δεν θα χρειαστεί να ψηφίσουμε πάνω σε αυτήν. Αυτά είναι τα σχόλια που έχω να κάνω εγώ επί των τροπολογιών. Που είναι λίγες σχετικά. Και νομίζω ότι είναι ένα σχετικά απλό θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Α, ο κύριος Στάλιν έχει δει στο λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις μονάχα. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ την κυρία Γένθεν για την πληρότητα της ε, παρουσίασής της για όλες αυτές τις, τις ε, απαλλαγές. Εγώ νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποιες ανταλλαγές απόψεων και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής για την πρόσκληση του Πατρική, ο οποίος ήρθε να μας παρουσιάσει τα θέματα του ΣΕΖΑΡ, γιατί έχουμε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Και επίσης υπάρχει το θέμα της ΙΑΣΑ. Όπως είπε η κυρία Γένσεν, οι τροπολογίες οι οποίες και έχουν κατατεθεί είναι γενικά πολύ καλές. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι που ισχύει για το ΣΕΡΑ. Αυτό όμως το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι δεν θέλω να υποστηρίξουμε καταρχήν όλες αυτές τις απαλλαγές. Αλλά όταν η κυρία Γένσεν έχει τονίσει τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, παραδείγματος χάρη στην Ιάσα και στο Σέζαρ, μπορούμε τώρα μετά από αυτά που μας είπε ο Πατρική για το Σέζαρ γιατί είναι ικανό άτομο και ξέρει περί τίνο πρόκειται. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι η βιομηχανία αυτή τη στιγμή επενδύει σημαντικά χρηματικά ποσά και στο, και στο ΣΥΖΑ και σε άλλες ενέργειες. Επομένως δεν είναι μοναχα θέμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΙΑΣΑ τα δύο τρίτα της χρηματοδότηση έρχεται από, την, από τον ιδιωτικό τομέα, από τη βιομηχανία. Μήπω μπορούν να σταματήσουν τα πηγαδάκια εδώ πέρα στην αίθουσα συνεδριάσεων, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Μερσή, κύριε Πρόεδρε. Άλλο είναι το να κάνουμε μια συζήτηση για το τι δίνουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λειτουργήσουν αυτοί οι φορείς. Αλλά τα δύο τρίτα για την ΙΑΣΑ έρχονται από τη βιομηχανία, οι οποίες δημιουργούν και θέσεις απασχόλησης. Επομένως όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερε και οι ελλείψεις που παρατηρούνται δεν είναι κάτι Θέλουμε να υποστηρίξουμε τη διαδικασία της απαλλαγής και να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα αυτά στο μέλλον και ορισμένε από τις τροπολογίες είναι πολύ θετικέ, αλλά παράλληλα χρειάζεται να έχουμε και την εξασφάλιση ότι θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα σημαντικά θέματα όταν δούμε το πόσα χρήματα διακυβεύονται και πόσο μεγάλη είναι η σημασία αυτών των αποκεντρωμένων φορέων. Νομίζω ότι θυμόσαστε κύριε Πρόεδρε ότι τονίσαμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε τους εκπροσώπους της ΙΑΣΑ εδώ γιατί πρέπει πράγματι να συζητήσουμε τα θέματα με αυτούς. Είπατε ναι εφόσον το συμφωνήσουν όλοι οι συντονιστές. Ελπίζω θα συμφωνήσουν οι συντονιστές και θα κάνουμε τότε κάτι τέτοιο. Σίγουρα θέλουμε να προχωρήσουμε και ενδιαμέσως θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Γέντσεν για το έργο της αλλά είμαστε κάπως εν Θα υποστηρίξουμε αυτές τις απαλλαγές με τα ερωτηματικά τα οποία τέθηκαν. Θέλουμε να ξέρουμε ότι τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα θα ληφθούν. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας διαβεβαιώσει, ίσως θα μας διαβεβαιώσουν οι αποκεντρωμένοι φορείς. Κάποιος πρέπει όμως να μας διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν αυτές οι απαραίτητες ενέργειες γιατί είναι δύσκολο το θέμα της απαλλαγής της ΙΑΣΑ και του ΣΕΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φώστερ ήταν πάρα πολύ διπλωματική στα σχόλια που έκανε. Εγώ όμως δεν θα είμαι τόσο πολύ. Γιατί βαρέθηκα πια με αυτή την Ιάσα. Βαρέθηκα λοιπόν με αυτή την Ιάσα πρώτον γιατί δεν μας δίνει καμία επιστροφή στα χρήματα που δίνουμε. Ε, και η κυρία Φώστερ μάλιστα αναφέρθηκε σε κάποια από τα ε, αρνητικά στοιχεία αλλά ε, λίγο με το γάντι εγώ πια έχω βαρεθεί να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και κύριε Πρόεδρε ξέρετε πολύ καλά ότι το τελευταίο προέρχεται από τη... από την Ένωση Ανεμοπτεριστών ε, και ε, ε, αυτός βεβαίως είναι, αυτή είναι ένας τομέας αναψυχής. δεν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί εδώ και εν πάση περιπτώσει άλλωστε έχει ήδη ρυθμιστεί ικανοποιητικά από μόνο το τομα, τομέας αυτός. κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα και να χάνω όλο και περισσότερο την ψυχραιμία μου όσο τα λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτή η Άσα θα πρέπει να μας αποδώσει λογαριασμούς ε, και ε, νομίζω ότι και μια ακρόαση του Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική για το θέμα αυτό. Δεν έχω ούτε εδώ εκπρόσωπο της Κομισιόν. Έφτασε η κυρία Γιάλα Σέντερς όμως. Εδώ είναι η έκθεσή σας, είσαστε και σκιώδης για το επόμενο, για το άλλο θέμα να τα ακούσετε όλα πρώτα τα σχόλια και μετά να απαντήσετε. Είχα πει δύο λόγια στην παρουσία της έκθεσής μου για τον οργανισμό των σιδηροδρόμων. Υπάρχει μονάχα ένα, μια, μια, ένα γραφείο στον σταθμό της ε, ΛΙΛ ε, και εν πάση περιπτώσει η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια μείωσης του κόστους. Ε, δηλαδή να υπάρχει ένα γραφείο μικρό στο οποίο να μπορούν να γίνονται συνεδριάσεις και να είναι κοντά στο hub αυτό, κοντά στον κόμβο, τον σιδηροδρομικό. Ε, και νομίζω ότι ε, με τα μισά χρήματα μπορούμε ε, να επενδύσουμε έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το 50% από τα αρχικώς προβλεπόμενα στον προπολογισμό. Στην πραγματικότητα όμως, εάν δούμε τα, τα στοιχεία ε, το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο αυτού του οργανισμού όσον αφορά ε, το, τα κτίρια είναι πολύ χαμηλότερο γιατί ακριβώς όπως σας εξήγησα προηγουμένως ε, υπάρχει ένας καταμερισμός των εξόδων ενοικίασης με άλλους οργανισμούς βέβαια αυτό δεν μπορεί να αλλάξει την ουσία της τροπολογία σας. Όμως να σας ξαναπώ ότι στο σιδηρόδρομο για τα θέματα δηλαδή σιδηροδρομικά πολύ δύσκολα βρίσκει κανείς ε, εμπειρογνώμονες. Ε, πρώτον γιατί το είδος που ασχολείται με μελέτες σιδηροδρομικές ε, μεγαλώνει, γυράσκει και από την άλλη πλευρά και από την άλλη πλευρά οι εθνικοί οργανισμοί και οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μας δίνουν τους εμπειρογνώμονες και επομένως δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να καλύψουμε αυτή την υποχρέωση. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, κυρία Γιάλα Σέντερ, να κάνετε και την παρουσία της εκθεσής σας και ε, εκεί που είστε σκιώδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Και συγγνώμη εγώ ήμουν για τον προπολογισμό και με τον Υπουργό τη Ισπανία συζητούσα και πρέπει να τρέξω από ένα σημείο, λίγο αυτό άργησα. Λοιπόν, η απαλλαγή λοιπόν για τι μεταφορέ τώρα. Υπάρχουν δύο τροπολογίε του κυρίου Κράμερ που βρίσκω μια χαρά. Η μία από τις δύο γιατί είναι μια ιστορική αναφορά και συμφωνώ. Και η δεύτερη διότι υπογραμμίζει, αιτιολογεί τέλο πάντων καλύτερα την ανάγκη να μπορούμε να εξηγούμε στους επιβάτες τα δικαιώματά τους. Οπότε συμφωνώ καταρχήν και με τις δύο. Αν συμφωνούν ε, και άλλοι με τη δικιά μου τροπολογία, πέντε που μιλάει για τον τουρισμό, υπογραμμίζει πιο ιδιαίτερα τον τουρισμό, ώστε να είναι παρόν στην απαλλαγή, κατά τα άλλο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα την έκθεση της κυρίας Γένσεν, που προσπάθησε να κοιτάξει όλους τους οργανισμούς που είναι σημαντικοί για μας. Για την ΕΜΣΑ έχω δύο τροπολογίες γιατί πιστεύω ότι πρέπει, είναι πολλά χρόνια τώρα που έχουμε την ΕΜΣΑ. Έχουμε συζητήσει χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Έχει αναγνωρίσει η τουλάχιστον ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία, το κόστος και την ασφάλεια ε, πρέπει να έχει λόγο. Αλλά θέλουμε και τα σχέδια και τις προβλέψεις. Ε, ναι, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει εδώ πέρα μια ασάφεια, όσον αφορά την χρήση των προβλέψεων και τις υποχρώσεις δηλαδή πληρωμών και τις πληρωμές αυτές καθ' αυτές. Δεν μας φαίνεται ξεκάθαρο το σύστημα, ενώ ο οργανισμός είναι πολύ σημαντικός. Οι τροπολογίες μου αυτό που θέλουν είναι να ενισχύσουν την απέτηση που έχουμε από τον οργανισμό για πιο ξεκάθαρους λογαριασμούς. Θέλω τώρα να ρωτήσω για τον Οργανισμό Ασφαλής της Αεροπορίας. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες και εδώ απαιτώντα πιο συγκεκριμένα σχέδια. Γιατί και η Κομισιόν μας έχει στείλει το μήνυμα ότι χρειάζεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Στις δύο τροπολογίες θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή της ομάδας εργασίας της διοργανικής για τους οργανισμούς ποια είναι. Είναι ο έλεγχος των διαδικασιών. Τότε ναι, να ενισχυθεί. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να ξεφύγει ο έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμού, ο έλεγχος των δημοσιονομικών και ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό του οργανισμού η ομάδα θέλω να ενισχύει τον έλεγχο αυτών. Τίποτα άλλο. Τέλος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Εδώ θέλω να πω ότι συμφωνώ, καταρχήν, μου το εξήγησε και ο κύριος Ρίκε πριν, το θέμα των δύο εδρών. Μπερδευόμαστε και μπερδεύουμε και τους πολίτες. Αυτό πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Να γίνει μια προσπάθεια λοιπόν από το κράτος όπου είναι γεγραμμένος οργανισμός, ώστε να βελτιωθεί η προβολή. Τέλος, για τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές, θέλουμε η κυρία Γένσεν που μιλάει για ε, δυσκολίες, μάλλον δεν λέει δυσκολίες εκείνη, μιλάει για ελλείψεις, εγώ θα προτιμούσα δυσκολίες. Πρέπει γρήγορα να αυξηθεί το προσωπικό. Να βρεθεί εδώ πέρα ένας συμβιβασμός καλύτερα. Ο κύριος Ρίκε αλλιώς έχει δίκιο ότι δεν πρόκειται για ελλείψεις, αλλά πρόκειται για μια αδυναμία που έχει ο οργανισμός να ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά. Κυρία Γέννησε, θέλετε να επανέλθετε όσο διπλωματικά όσο η κυρία Φώστερ και όχι με τόσο μεγάλη οργή όπως ο κύριος Μπράτβερν. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Συμφωνώ πλήρως με την κυρία Φώστερ γιατί είναι θετικό η Επιτροπή μας να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους των αποκεντρωμένων φορέων και ιδίως της ΙΑΣΑ για να συζητήσει τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε εμείς, τα προβλήματα τα οποία βλέπουν αυτοί, ενώπιση του μέλλοντος. Αναφερθήκατε σε αυτή την διαθεσμική ομάδα. Δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα λόγω του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι αποκεντρωμένοι φορείς δημιουργούνται ρυθμιστικού χαρακτήρα. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικαθιστούν κάποιες υφιστάμενες αρχές, αλλά όλα αυτά είναι από προϋπολογισμούς που είναι από τμήμα του προϋπολογισμού που είναι εκτός των διοικητικών δαπανών. Είναι σαν να κλέβουν τα λεφτά μας που είναι λεφτά για λειτουργικές δαπάνες για να, κάνουν, για να καλύψουν διοικητικές δαπάνες. Αυτό θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι κάνουν αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο έχει χωρίσει σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν ότι όταν δημιουργείται ένας αποκεντρωμένος φορέας θα πρέπει να υπάρχει μια πάγια διαδικασία για την αντιμετώπιση της, να υπάρχει μια μελέτη αντικτύπου, να υπάρχει πλήρης αξιολόγηση του κόστους και της ωφέλειας της δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου φορέα και πριν από δύο χρόνια η Κομισιόν μας παρουσίασε μια αξιολόγηση του σύνολου συστήματος και είπε ότι πρέπει να κάνουμε ρεκτιφιές στο σύστημα, να το τροποποιήσουμε και να έχουμε και μια νέα διαθεσμική συμφωνία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η διαθεσμική ομάδα εργασίας. Θα πρέπει να δούμε τώρα ποιοι επίτροποι θα συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα, αλλά πριν από τις εκλογές ήταν ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, ο Επίτροπος για τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού, τρεις βουλευτές επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιος κόσμος από το Συμβούλιο. Τώρα έχουμε εκπροσώπους από τις έξι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες και φυσικά και εγώ είμαι μέλος αυτής της διαθεσμικής ομάδος και προχωρούμε σε πολλές μελέτες για το πώς λειτουργεί το σύστημα των αποκεντρωμένων φορέων, πώς εξελίσσεται και ποια είναι τα κοινά προβλήματα τα οποία βλέπουμε και ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Ο στόχος μου δεν είναι να αντικαταστήσω την Επιτροπή μας ή την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ή την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όχι. Είναι απλώς μία εξέταση όλων των προβλημάτων ώστε να προχωρήσουμε προς μια νέα διαθεσμική συμφωνία. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και να εξετάσουμε την ουσία στο τωρινό πλαίσιο αλλά συγχρόνως να έχουμε και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια πιο πολύ εκβάθρων μεταρρύθμισης. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι κοινά σε πολλούς αποκεντρωμένους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη ο κανονισμός υπηρεσικής κατάστασης που δεν έχει πάντα νόημα για αυτούς τους μικρούς φορείς, οι δημοσιονομικοί κανονισμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα. Θυμάμαι ένα φορέα αποκεντρωμένο που μας είπε ότι είναι αδύνατον να έχουμε κάποια απάντηση σε μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 30 κινητά τηλέφωνα υπάρχει και μια σειρά πιο θεμελιωδών προβλημάτων ότι υπάρχει ένα ευρύ διοικητικό συμβούλιο με εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν έχει και αυτή ένα ρόλο, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος έχει την πραγματική ευθύνη. Θυμάμαι που είχα θέσει ένα ερώτημα στον κύριο Μπαρό, που ήταν τότε ο Επίτροπος Μεταφορών, για ένα ζήτημα που αφορούσε κάποια αεροσκάφη τύπου DAS 8 ή κάτι τέτοιο, τα οποία δεν επέτρεπαν να πετάνε η Αυστρία και η Δανία, ενώ η Άσα τα άφηνε να πετάνε ελευθέρως και μεγάλη χαρά. Και ρώτησα τον Επίτροπο τι είναι αυτό το πράγμα. Η Άσα δουλεύει για την Μπομπαρτιέ ή οι εθνικές υπηρεσίες κάνουν κάτι λάθος στον έλεγχο των αεροσκαφών αυτών. Και είχε μεγάλη δυσκολία ο κύριος ε, Μπαρό τότε να αντιμετωπίσει τα δικά μου ερωτήματα, τα ερωτήματα του κύριου Λάιχτφριντ και άλλων και έβλεπα στο πρόσωπό του ότι δεν του άρεσε ο τρόπος που το αντιμετωπίζαμε αυτό γιατί όλοι αυτόν κατηγορούν Όλοι επιτίθενται εναντίον του, αλλά αυτός δεν μπορούσε να πει εντάξει θα απολύσω το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα αυτού. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού βρίσκεται η τελική ευθύνη σε όλους αυτούς τους αποκεντρωμένους φορείς. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο αυτό που κάνει η διαθεσμική ομάδα και πρέπει να κάνουμε το ίδιο εγχείρημα και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό θα είναι ένα επαναλαμβανόμενο εγχείρημα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, υποστήριζω τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει και θα ξαναδώ και πάλι την τροπολογία του κυρίου Λουίκη σε σχέση με το προσωπικό. Και γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τη σωστή στελέχωση για την ΕΡΑ για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμου. Έχουμε εμπειρογνώμονε για εθνικού σιδηροδρόμου, αλλά όχι για Ευρωπαϊκού σύνδρομου. Κύριε Κούν, θέλετε να λάβετε το λόγο, εν συντομία. Δυστυχώ ο συνάδελφό μα ο κύριο Ήταλα, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά όλοι είχαμε προβλήματα με τι ε, συνθήκε μεταφορών σήμερα. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γένσεν για τον Ευρωπαϊκό Φορέα ε, Μεταφορών Διασυνδρόμου. Ο κ. Ρικέ έχει πολύ καλές προτάσεις, οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε για την αξιολόγηση της Κομισιόν έχω μία ε, αίτηση, μία παράκληση και αναφέρομαι στην κυρία Αγιάλα Σέντερ, πρόκειται για την τροπολογία 2, παράγραφος 9α. Εκεί θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα μέχρι τον τομέα του τουρισμού και το δεύτερο χαιρετίζει τις νέες νομικές κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μια χωριστή ψηφοφορία στο σημείο αυτό. Πάντα μπορείτε να το ζητήσετε κύριε Κούν. Εφόσον μας το έχετε πει εγκαίρως ότι θέλετε χωριστή ψηφοφορία, Πάντα μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αν τώρα συμφωνεί η κυρία Αιάλα Σέντερ με αυτό, είναι διαφορετικό. Αλλά πάντα μπορείτε να ζητήσετε χωριστή ψηφοφορία. Ινιές. Ναι. Μια στιγμή κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα ήταν μέχρι πού φτάνει αυτή η χωριστή ψηφοφορία. Φτάνει μέχρι την τελευταία γραμμή που υποστηρίζονται από ένα πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Παράγραφος 9α, λέει ο κύριο Κούν, εντάξει. Η τροπολογία 2. Το πρώτο τμήμα λοιπόν θα πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί που λέει ο τομέας του τουρισμού. Το δεύτερο τμήμα στη συνέχεια και, χαρακτη... και χαιρετίζει το νέο νομικό κτλ. Εντάξει. We have now not uh, the voting situation. But we would assume that if you want to Εάν θέλετε να κάνετε χωριστή ψηφοφορία, θεωρούμε ότι δεν συμφωνείτε με ένα από τα δύο τμήματα. Αν θέλετε λοιπόν χωριστή ψηφοφορία, το καταγράφει η γραμματεία, θα το κάνουμε και θα δούμε τι θα προκύψει από την ψηφοφορία. Εντάξει, δικαίωμά σα είναι προφανώ να ζητήσετε ω πολιτική ομάδα μια χωριστή ψηφοφορία. Εντάξει, πάμε στο επόμενο θέμα. Η έκθεση του κυρίου Ελ Χαντραουί. Ο κύριος Ελ Χαντραουί είναι τώρα όμως στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων όπου αντιμετωπίζει μια άλλη έκθεση. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως τη συζήτηση για τις του. Θα ήθελα εκ μέρους του κυρίου Χαντραουή να κάνω μια γενική παρουσίαση και μπορεί να προσθέσει διάφορα σημεία όταν επανέλθει. Νομίζω το κύριο θέμα το επίμαχο εδώ είναι η συμπερίληψη ανεξαρτήτων αυτοαπασχολούμενων οδηγών στους κανόνες για το χρόνο εργασίας Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ήταν λίγο χωρισμένο όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, το πήρε μία ομάδα, μετά το έδωσε σε μία άλλη ομάδα κτλ. Ε, βλέπουμε εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός όσον αφορά την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ο κύριος Αλχαντράουι προσπάθησε να βρει μια συμβιβαστική λύση συμπεριλαμβάνοντας ε, τους αυτοαπασχολούμενους ε, οδηγούς και ξέρω ότι προτείνει να ε, λαμβάνονται ε, υπόψη και οι ώρες φορτοεκφόρτωσης μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό πέρασε από την Επιτροπή γιατί, ή θα περάσει γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο βασίστηκε σε πολύ μεγάλη συζήτηση επί της οποίας δεν υπήρξε συμφωνία. Ξέρω ότι ο κύριος Κρός και νομίζω ότι και η κυρία Γένσεν έχουν ε, υπογράψει κάποιες τροπολογίες βλέποντας το θέμα από τελείως διαφορετική πλευρά. Ε, δηλαδή λένε ότι θα πρέπει ε, να συμπεριληφθούν οι οδηγοί φορτηγών ε, και κάτω από 3,5 τόνους. Ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι θέλουν ε, να εφαρμοστούν για αυτούς τους οδηγούς, δηλαδή και για κάτω από, 3,5 τόνους ε, και οι οδηγίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ε, και Νομίζω ότι ούτε από αυτού υπάρχει μεγάλη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γίνει συζήτηση όσον αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Βλέποντας απ' έξω ε, ε, το κείμενο αυτό, εάν εγκριθεί η γραμμή του εισηγητού στην Επιτροπή Μεταφορών, ενδεχομένως θα μπορέσει να αποτελέσει βάση μια συμβιβαστική λύσης στην Επιτροπή Απασχόλησης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν στοιχεία της έκθεσης τα οποία μπορούν ε, να καταλήξουν ε, στην ε, περιοχή της απασχόλησης, της Επιτροπής Απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί δίνοντας την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για το θέμα αυτό. Λοιπόν, Σαΐντ, εγώ μέχρι τώρα έδωσα μια γενική έποψη, περιγραφή αν θέλει των ζητημάτων που συνδέονται με το θέμα αυτό. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, περίμενα να έρθεις, ε, να αναλάβεις εσύ τώρα. Λοιπόν, ε, έδωσα κάποιες γενικές αρχές. Ε, εσύ θα μας πεις λεπτομέρειες και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Βέβαια δεν είναι καλή ιδέα να παρουσιάζει κανεί συγχρόνω δύο εκθέσει σε δύο διαφορετικέ κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, αλλά τι να κάνουμε, μερικέ φορέ χρειάζεται. Εγώ θα υπογραμμίσω εδώ τι γίνεται με τις τροπολογίες. Έχουμε συζητήσει και με τους συναδέρφους, τους κοιόδης εισηγητές. Γενικά μιλώντας θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε με τις αρχές της έκθεσης, οι τροπολογίες συμφωνούν με τις αρχές της έκθεσης. Ξέρετε ότι προσπάθησα, έκανα μια απόπειρα να απομακρυνθούμε από το 50%-50% για τους αυτοπασχολούμενους και όχι. Έχω προτείνει κάποιες τροπολογίες, πάντως ξανά, που μιλάει για μείωση του διοικητικού άχθους και όπου λέω για παράδειγμα ότι για τους αυτοαπασχολούμενους η καταγραφή στο Μητρό πρέπει να είναι περιορισμένη. Να μην έχει δηλαδή ιδιαίτερο διοικητικό άχθος, αναφέρομαι εδώ και σε κάποια κριτήρια. Στην τροπολογία μου 32 λέει ότι για την κατηγορία αυτοπασχολούμενη είναι οι οδηγοί οι οποίοι δεν είναι αυτοί που κάνουν τις ε, συνεννοήσεις για τα ταξίδια και για το θέμα της περίοδου ανάπαυσης μιλάμε για τον ταχυγράφο και βάζουμε εδώ και την περίοδο φόρτωση-εκφόρτωσης. Και μιλάμε για ένα καταποκοπή χρόνο όσον αφορά τα καθήκοντα των αυτοαποσχολούμενων κατά το χρόνο εργασίας τους. Επίσης, αναφέρομαι και στα δεδομένα τα οποία καταγράφονται από τον ταχυγράφο. Είναι μερικά πράγματα που συνάδουν με τη γενική αντιμετώπιση. Υπάρχει πάντως αυτή η βασική αρχή που μας κάνει να μην συμφωνούμε για τον ορισμό της έννοιας. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αύριο θα ψηφίσουμε και θα δούμε τελικά ποια είναι η γνώμη της πλειοψηφίας της Επιτροπής αυτής. Και στην Ολομέλεια φυσικά πάλι θα διευκρινιστεί το θέμα. Αυτό σημαίνει τώρα για τις τροπολογίες των συναδέρφων συνάδελφος Γκρό και άλλοι έχουν υποβάλει διάφορες τροπολογίες. Μερικές από αυτές μπορώ να τις υποστηρίξω. Υπάρχει για παράδειγμα η πρόταση για τους de facto οδηγούς κάτω από 3,5 τόνους, να μην συμπεριληφθούν. Η δικιά μου ιδέα στην τροπολογία μου 27 ήταν ότι πρέπει να το δούμε αυτό πιο πολύ. Στην πράξη δεν είναι τόσο απλό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα φέρω δυσκολίες. Θα δούμε τι θα κάνει και το Συμβούλιο ε, και τι θα γίνει και στην ε, ε, Ολομέλεια και στο Συμβούλιο. Για μένα πάντως ο ορισμός των αυτοπασχολούμενων είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και στις δικές μου τροπολογίες, μεταξύ άλλων στη 30, θέλω να ακολουθήσω την ε, ίδια γραμμή που λέει ότι η έλεγχη πρέπει να είναι εθνική. Έχω κάνει κάποιες προτάσεις σχετικά με τους ελέγχους, αν πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι. Πάντως, το αν συμπεριλαμβάνονται και αυτοαπασχολούμενοι όχι είναι το κύριο πρόβλημα. Στην 31, δεν έχω πρόβλημα με τη συνέχεια της οδηγίας. Για την κυρία Φορμανκόλ, που λέει εντάξει είναι καλή ιδέα. Αν είναι τα κράτη-μέλη, τότε εκεί να εντοπίζουν ποιοι είναι οι ψεύδο αυτοαπασχολούμενοι. Τέλος, τροπολογία Λίχτεμπερκ. την στηρίζω όσον αφορά τη νυχτερινή περίοδο. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε. Αυτές είναι κάποιες παρατηρήσεις που είχα να κάνω με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε ομιλητές εγώ προς το παρόν. Αν μπορούμε να μείνουμε στα δύο ή τρία λεπτά τον καθένα. Ξέρω ότι είναι σημαντικό το θέμα αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα όπου δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας παρά μόνο με ψηφοφορία. Ξεκινάμε τον κύριο Κούν από το ΕΛΚ. εκ μέρους του ΕΛΚ. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι δικές μας τροπολογίες 19 και 30 του κύριου Γκρό είναι πολύ σημαντικές. Θέλουμε εδώ να τονίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε σε μια συμβαστική λύση και τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων τα οποία τα οδηγούν εργαζόμενοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Έχουμε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ακριβώς τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται στον τομέα των οχημάτων μέχρι τριών και μισού τόνου. Αν θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τα πράγματα θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα αυτό. Δεν συμφωνούμε όλοι οι ανεξάρτητοι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί να μπουν στην σφαίρα εφαρμογής της οδηγίας για το χρόνο εργασίας και μας φαίνεται επίσης το θέμα της γιαλαντζή ε, ανεξαρτησίας των οδηγών αυτών, αυτών που είναι ψεύδο αυτό απασχολούμενοι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά πιστεύουμε και επίσης ο ορισμός της νυχτερινής εργασίας έχει καθοριστεί ήδη σε προηγούμενες οδηγίες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια νέα διατύπωση και θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα το ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μονάχα οι ασφάλειες στους δρόμους, θα πρέπει να μας, να μας απασχολήσουν επίσης και τα κοινωνικά στοιχεία της απασχόλησης αυτής. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει μια πλήρης επανεξιολόγηση αυτής της οδηγίας μετά από δύο χρόνια για να δούμε κατά πόσον οδηγεί στα σωστά αποτελέσματα. Και για αύριο έχω μάθει από την κυρία ε, Γένσεν και τον κύριο Γκρός ότι για την 19 και για το 30 θα τεθούν ε, προφορικές τροπολογίες από το ΕΛΚ. Απλώς θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν δεκτές αυτές οι προφορικές τροπολογίες από τη μεριά του κόμματός μας. Σας λέω και πάλι ότι μπορούν να καταθεθούν τροπολογίες προφορικές εκείνη τη στιγμή, αλλά αν υπάρχει κάποια αντίρρηση προφανώς δεν θα γίνουν δεκτές. Έτσι λένε οι κανόνες. Κυρία Γέντσεν για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω βεβαίως τον εισηγητή για τις προσπάθειές του να φτάσει σε συμφωνία, αλλά νομίζω ότι εδώ είμαστε πειρασμένοι 50-50. Μπορώ να πω ότι οι τροπολογίες που υπέβαλα μαζί με τον κύριο Γκρός προσπαθούν να υπογραμμίσουν αυτά τα σημεία, αλλά να δώσουν και μία λίγο διαφορετική προσέγγιση, να προσεγγίσουν δηλαδή τα, τις ανησυχίες λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει εδώ να καλύπτουμε τους εν εργανομένους αλλά όχι ε, αλλά να καλυφθούν και από την ε, οδηγία για τον χρόνο εργασίας όπως και η οδηγή ταξί ας πούμε. Ε, κύριε Καντράου, εγώ θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει τέτοια αναφορά εδώ. Γι' αυτό υποβάλλαμε και τις τροπολογίες. Βεβαίως είναι περίπλοκο το ζήτημα και κατά κάποιο τρόπο υποχρεώθηκα να υποβάλω προφορική τροπολογία επί των άρθρων 19 και 30 όπου το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούμε αυτούς που δεν καλύπτονται από τις όρες οδήγησης και ανάπαυσης. Αλλά σε αυτήν την οδηγία υπάρχουν πολλές ε, ε, εξαιρέσεις που δεν ε, ε, καλύπτονται από την ε, οδηγία για τις ε, ώρες εργασίας Why we need, στρατιωτικά οχήματα κλπ. Ας πούμε η τροπολογία επί της 19 θα πρέπει να λέει κάπου στη μέση υπό το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας με ε, εξαίρεση για τους 3,5 τόνους. Ε, θα το συζητήσουμε όμως ξανά να δούμε έτσι ώστε να υποβληθεί κάτι σωστό. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε με την τροπολογία 27. Δεν συμφωνούμε όμως ε, ότι θα πρέπει να καλύπτονται και οι 3,5 τόνοι από ε, την ε, ε, οδηγία για την οδήγηση και την εργασία. Αυτά. Νομίζω ότι στο τέλος τη ψηφοφορία ε, θα έχει τραβήξει ο καθένα το δρόμο του. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γένσεν, θα ήταν καλό να ξεχωρίσουμε το χρόνο εργασίας και τον χρόνο οδήγησης. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το ίδιο άτομο μπορεί να κουραστεί είτε από την εργασία είτε από την οδήγηση. Και αυτό σημαίνει ότι και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρξει πρόβλημα για την οδική ασφάλεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίσουμε την συνολική εργασία από το χρόνο οδήγηση. Ένα δεύτερο σημείο. Για τα άτομα τα οποία είναι φαινομενικά μονάχα αυτοαπασχολούμενοι, εκεί έχουμε τα πιο μεγάλα προβλήματα. Είναι σαφές και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται όπως θέλει εφόσον δεν δημιουργεί κίνδυνο για τον εαυτό του. Αλλά εδώ δεν είναι το πράγμα τόσο απλό. Γιατί είναι πράγματι πολύ μεγαλύτερο ο κίνδυνο από ένα κουρασμένο οδηγό όταν οδηγεί ένα πιο βαρύ όχημα. Βέβαια για τους 3,5 τόνους είναι προβληματικά τα πράγματα γιατί και ένα όχημα 3,5 τόνων μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές. Και δεν είναι σωστό να πούμε ότι κυκλοφορούν μονάχα σε μικρές αποστάσεις. Αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιες χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά δεν ισχύει στο κέντρο της Ευρώπης, στις κεντρικές περιοχές της Ευρώπης. Ακριβώς γιατί αυτός ο τομέας δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις, χρησιμοποιούνται πολύ τα μικρά αυτά οχήματα, τα οποία επομένως μπορούν να οδηγήσουν σε ιδιαίτερους κινδύνους. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε αυτή την παράκαμψη των κανόνων και να αγνοήσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με, τους, με τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Και έχετε δίκιο γενικά, είναι πολύ δύσκολο γενικά να ελέγξουμε ποιος είναι πραγματικά ανεξάρτητος και ποιος είναι μονάχα φαινομενικά ε, ανεξάρτητος, γιατί για να το πω με επιήχεια... η φαντασία και η δημιουργικότητα σε αυτό το τομέα είναι ανεξάντλητη. Αν θέλουμε εμείς λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ε, ισότητα ανταγωνισμού μεταξύ των λογικών ε, εργοδοτών και αυτών οι οποίοι οδηγούν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και συγχρόνως να προστατεύσουμε την ασφάλεια της ε, κυκλοφορίας και των οδικών μεταφορών θα πρέπει να πάρουμε μια σωστή απόφαση στον τομέα αυτό. Ο καθένα βέβαια τα βλέπει τα πράγματα σε αυτά τα θέματα από τη δική του οπτική γωνία. Για μένα όμω το πιο σημαντικό, όπως τόνισε πολύ καλά ο κύριος Ελκατράουε, είναι ότι εάν συνεχίσουν οι, οι ρήτρε αυτές να την χάνουν τόσο λίγο ελέγχου και στο μέλλον όπως γίνεται σήμερα, τότε και οι καλύτερε προδιαγραφέ δεν ωφέλουν σε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στον έλεγχο και στην αστυνόμευση. Ο κύριος Φαντάλεν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Έλγα Αντρά. Ξέρω ότι έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αλλά στην πολιτική πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Και τα είπαμε αυτά και στο Στρασβούργο. Εμείς έχουμε μια εντελώ διαφορετική θέση στο θέμα αυτό. Και αύριο θα το καταλάβετε στην ψηφοφορία ποια θέση της ε, ομάδας μου. Για τις τροπολογίες 24-25. Κάντε και Κόλ. Εδώ θέλουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Επίσης, για την προσπάθεια συμβιβασμού. Δεν ξέρω ακριβώς τελικά κύριε Κούν που είναι ο συμβιβασμός. Εγώ δεν τον βλέπω. Και αυτό που είπατε στα γερμανικά compromise bereit» εγώ δεν το βλέπω. Πραγματικά. Αλλά ελπίζω αύριο στην ψηφοφορία να ξεκαθαριστούν λίγο περισσότερο τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, να κάνω μια Όσοι θέλουν ε, κατά τμήματα ψηφοφορία να ενημερώσουν τη γραμματεία, να το ξέρει και έτσι να είμαστε έτοιμοι αύριο για την ψηφοφορία, να μην δυσκολευτούμε παραπάνω. Κύριε Μπράτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, και σύμφωνα με τα σχόλια τα δικά σας ε, ε, και λαμβάνοντας υπόψη και ότι οι τροπολογίες χωρίζονται στην ουσία σε τρεις ομάδες δείχνει ότι δεν έχουμε σύμπνοια όσον αφορά το θέμα αυτό. Το πρώτο ζήτημα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι. Θα θυμάστε φαντάζομαι ότι από την αρχή εγώ είχα πει ότι στην δικιά μου εκλογική περιφέρεια στην οποία υπάρχουν περίπου 900 ε, διαφόρων μεγεθών εταιρείες που ασχολούνται ε, με αυτού του είδους ε, το θέμα και είπα ότι τουλάχιστον οι μικρές εταιρείες πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο και τα προβλήματα που τους δημιουργεί. Δεύτερον, ε, αναφερθήκατε στον φορτηγατζή το φορτηγατζί με, το, με τα, τη γνωστή φιγούρα αυτή με το μικρό φορτηγάκι. Ε, εγώ νομίζω σχετικά με το αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι. Ε, ε, να σας πω από τη δικιά μου περιφέρεια. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ε, πολλά μικρά τέτοια φορτηγάκια γιατί ακριβώς έχουμε πολλές ε, αγροτικές περιοχές. Ε, πρόκειται για φορτηγά τα οποία μεταφέρουν πράγματα σε απομακρυσμένες φάρμες, σε απομακρυσμένες περιοχές. Δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να μπουν τέτοιου είδους φορτηγά εδώ. Βεβαίως το πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως στην Αυστρία το καταλαβαίνουμε αλλά δεν μοιάζει ταιριάζει καθόλου με το ζήτημα, ε, το πρόγραμμα που παρουσιάζεται ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και ακριβώς σε αυτή την περίπτωση ο καθένας θέλει το δικό του κουστούμι. Δεν υπάρχει ένα μέγεθος κουστούμιου που να πηγαίνει σε όλους. Τρίτο, το θέμα του ορισμού της νυχτερινής εργασίας. Μέχρι τώρα τουλάχιστον ε, η αντίληψη που είχαμε ήταν ότι η νυχτερινή εργασία είναι θέμα επικουρικότητας και επομένως θα πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη τι θα ορίσουν νυχτερινή οδήγηση, νυχτερινό οδηγό κτλ. Ε, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να οδηγηθούμε σε αυτό το σφάλμα. Είναι λάθος ο δρόμος που ακολουθούμε και για αυτό το θέμα. Εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω ε, οτιδήποτε το οποίο θα πάρει από, την, από τα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων την δυνατότητα να αποφασίζουν τι είναι ε, νυχτερινή οδήγηση και να το δώσει στην Κομισιόν. Ο κύριος Πασκαρέλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση έκανε μια, ε, η, η Επιτροπή έκανε μια πρόταση με την οποία δεν αλλάζει. Ε, α, κύριε Πασχαρή, δεν έχουν τελειώσει... Δεν, ε, δεν θέλ, ε, γίνονται κάποιες συζητήσεις, πρέπει να σταματήσουν αυτές. Ναι, ναι, ναι, ναι δεν κατάλαβα στην αρχή τι λέγατε. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση ως Κομισιόν, δεν την αλλάζουμε. Όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι το μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ε, ακριβώς ε, η προστασία των εργαζομένων, η υγεία των εργαζομένων και η υγιεινή τους στη θέση εργασίας τους. Αλλά δεν νομίζω ότι εδώ είναι το κατάλληλο μέρος για να ασχοληθούμε με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κ. Κατράουη έκανε μια προσπάθεια να βρει συμβαστικές λύσεις. Βλέπω όμως ότι και στην Επιτροπή σας ε, και στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, που ήμουνα ε, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αμφισημία όσον αφορά τις θέσεις των διαφόρων πλευρών και εν πάση περιπτώσει θα γίνει η ψηφοφορία και θα δούμε. Εμείς έχουμε τη δικιά μας θέση, έχουμε τις δικές μας απόψεις όσον αφορά ορισμένε τροπολογίες εμείς θα θέλαμε ε, να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμφωνία επου, επί του κειμένου. Ε, βλέπουμε όμως τροπολογίες 1, 6, 7, 10, 22, 29, 32, 37, 40 οι οποίες ε, διαρκώς συμπεριλαμβάνουν την έννοια του αυτοαποσχολούμενου οδηγού δεν μπορούν να τύχουν τις εύνοια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δεν είναι ε, δυνατόν ε, να ε, μπουν, να αλλάξουν κάποια κατηγορία χωρίς να, τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση για περαιτέρω γραφειοκρατικό διοικητικό άχθος. Ε, απ' την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν εμείς να κατεβούμε σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειες όσον αφορά τους κανονισμούς. νομίζω ότι Εάν ε, οδηγηθούμε προς τα εκεί θα έχουμε τελικά ε, νομοθετικές πράξεις οι οποίες πάρα πολύ δύσκολα αν όχι αδύνατα ε, θα μπουν σε λειτουργία και θα τεθούν σε ισχύ. Κοιτάξτε, έχουμε έναν γενικό κανόνα που λέει ότι η αυτού του είδους οι κανονισμοί αφορούν τα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε ε, ad hoc σε μία ε, συγκεκριμένη περίπτωση την, ε, ε, την κατηγορία, την αφορούμενη κατηγορία. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μόνο για αυτό το ζήτημα ε, θα συμπεριλάβουμε και φορτηγά κάτω από 3,5 τόνους. Κοιτάξτε, έχουν γίνει μελέτες όσον αφορά το ενδεχόμενο εφαρμογής όλης, όλων των κανονιστικών ρυθμίσεων για τις μεταφορές στα φορτηγά κάτω από 3,5 τόνους. Για την ώρα δεν έχουμε οδηγηθεί σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα ότι θα πρέπει να κάνουμε κάνουμε κάτι τέτοιο, διεύρυνση δηλαδή του πεδίου εφαρμογή. Ούτε όμως μπορούμε ε, αναπερίπτωση να τροποποιούμε το πεδίο εφαρμογήσε των ε, οδηγιών. Απ' την άλλη πλευρά, όλες οι τροπολογίε οι οποίες αποσκοπούν σε, καλύτερη ε, και σε καλύτερο και σαφέστερο ορισμό ε, των ε, εργαζομένων και που αποσκοπούν σε καλύτερη προστασία των εργαζομένων βάσει τη εφιστάμενης και ισχύουσα νομοθεσίας μας βρίσκουν σύμφωνους. Μπορούμε να, ψηφ... να ε, στηρίξουμε λοιπόν όλες αυτές ε, τις ε, τροπολογίες οι οποίες περαιτέρω διευκρινίζουν τις βασικές αρχές. 20, Βόρτμαν Κόλ, η πρώτη τροπολογία του κυρίου Χαντράουι, η τροπολογία της κυρίας Σικάου σχετικά με το να ευαισθητοποιηθούν όλοι όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ψηφοφορία αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομα, Σαΐντ, για να ξεκινήσουμε και με τους συντονιστές. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχετε ήδη άποψη προς τη μία κατεύθυνση, δεν πρόκειται να πιστείτε τώρα, οπότε σύντομα. Ε, αυτό είναι δημοκρατία στο κάτω-κάτω. Μα είμαστε μέσα στα χρονικά Έχουμε τρία λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, λέει ο κύριος Αλκατραουή. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τόσα μας είπε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Στην παλιά οδηγία νομικά μιλώντας, δεσμευόμαστε. Οι αυτοπασχολούμενοι συμπεριλαμβάνονται. Αυτή είναι πραγματικότητα. Οπότε ό,τι παρατηρήσεις γίνονται, ότι μα δεν είναι λογικό, δεν είναι ελεγχόμενο, δηλαδή δεν μπορεί να, γίνει, να γίνονται καλά έλεγχοι κτλ. Μπορούμε να τα πούμε, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε έτσι γιατί ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα σε αυτό. Τώρα, για τους ελέγχους πιο συγκεκριμένα. Όντως, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ακριβώ γι' αυτό και έκανα την προσπάθεια να προσπαθήσω να εξευρωπαίσω κάπως τους ελέγχους. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Σιγά σιγά μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση και σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, η έλεγχη είναι ένα περίπλοκο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το σκεφτεί, να οριμάσει δηλαδή η ιδέα και να μας κάνει μια πρόταση. Βέβαια κατάλαβα ότι δεν την ενδιαφέρει την Επιτροπή κάτι τέτοιο, ίσως έχει πολλή δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχει η Επιτροπή. Αλλά θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία 19